σχετικά με, την, με το τελευταία στιγμή επανασυνδέθηκε το θέμα σας των διμερών σχέσεων με την Τουρκία ε, και με το θέμα της διένεξης στον Αγκόρνο Καραμπάχ και με τους Τούρκους αδερφούς του Αζερβαϊτζάν. Είναι παράλογο κατά την γνώμη μου και είναι αντίστοιχο της, το, να κλείνει η Ελλάδα τα σύνορά της προς την Τουρκία σε αλληλεγγύη με τους Ελληνοκυπρίους. Δεν μπορούν να, να κρατούν ε, τα σύνορα κάποιοι κλειστοί εν ώψη διεθνών ε, διανέξεων η Αρμενία δυστυχώ στηρίχθηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα στη ρωσική στρατιωτική προστασία και είναι τραγικό το ότι η γενοκτονία του 1915 δεν ε, έχει τύχει επαρκούς ε, σημασίες από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα θέλαμε να υπάρχει διαφοροποίηση στην Αρμενία και να ε, υπάρξουν ενισχυμένε οικονομικές σχέσεις, ούτως ώστε να υποφεληθεί η Αρμενία. Κύριε Πρόεδρε, έχετε πολλούς φίλους, θέλω να το πιστέψετε αυτό στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μπορείτε να στηρίζεστε στη δική μας υποστήριξη. Είμαστε κατά οποιασδήποτε στρατιωτικής λύση στη διένεξη, στην παγωμένη αυτή διένεξη ένταξη στο Ναγκόρνο Καραμπάχ και θα ήθελα να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου για τον πρόσφατο θάνατο έξι στρατιωτών σε αυτή τη διένεξη, στρατιωτών και από την Αρμενία και από το Αζερβαϊτζάν. Ε, και διαφωνούμε με τις δηλώσεις ε, του ε, Προέδρου Αλίγεφ που πιστεύει ότι τα πετροδολάρια μπορέσουν να αποτελέσουν μια λύση για αυτό το θέμα. Υποστηρίζουμε πλήρως την γενευτική διαδικασία μέσω της ομάδας Μίνσκ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Είμαι εσύ που είναι η μόνη λέξη που γνωρίζω στα αρμενικά. Ευχαριστούμε κύριε Τάνοκ. κύριε Φιγκινού. Τα δύο Ευχαριστώ ε, κύριε Πρόεδρε, κυρία Βραχανιάν. Εκ μέρου τη ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών θα ήθελα να σα καλωσορίσω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι η πρώτη σα επίσκεψη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ελπίζω ότι θα έχετε θετικέ εντυπώσει από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από του Ευρωβουλευτέ και ελπίζουμε ότι θα συνεργαστούμε πιο στενά στο μέλλον. Με μεγάλη μου χαρά είδα ότι σε, μια, σε ένα πολύ δύσκολο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον Διεθνώ, η Αρμενία παραμένει σε σταθερό επίπεδο, προσπαθεί να επιτύχει μεταρρυθμίσεις, ακόμη και αν αυτέ οι μεταρρυθμίσεις δεν έχουν το ρυθμό που εμεί θα επιθυμούσαμε, Πάντω ακολουθεί θετική κατεύθυνση και στις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, χαίρομαι που άκουσα ότι είπατε ότι αξιολογείτε θετικά την πρωτοβουλία τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την ανατολική εταιρική σχέση. Αυτό θα είναι προς όφελος των διμερών σχέσεών μα αλλά και θα βελτιώσει βελτιώσει το πολυμερές ε, πλαίσιο με τις έξι χώρες που συμμετέχουν στην ανατολική αυτή η εταιρική σχέση. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι η περιφερειακή συνεργασία και οι καλές ε, σχέσεις γειτονία, αυτή η πολυμερής προσέγγιση, είναι κάτι πολύ σημαντικό για οποιαδήποτε χώρα που επιθυμεί να προσεγγίσει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αν μου επιτρέπετε να κάνω ένα σχόλιο και για την έκθεση για τη στρατηγική στο Νότιο Κάφκασο. Πιστεύω ότι το πιο σημαντικό σημείο στην έκθεση αυτή είναι ότι με μεγάλη πλειοψηφία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να δείξει μεγαλύτερη δραστηριότητα και να αναπτύξει μια στρατηγική για το Νότιο Κάφκασο. Το πώ θα διαμορφωθεί αυτή η στρατηγική θα εξαρτηθεί και από το διάλογο που θα έχουμε μαζί σα και με τι άλλε δύο χώρε τη ε, περιφέρεια. Έχω μια ερώτηση. Εκτός από το προφανές ε, γνωστό ζήτημα της διένεξης των Αγκόρνο Καραμπάχ, θα ήθελα να σας ρωτήσω πού βλέπετε εσείς τις βασικές απειλές για την θετική ανάπτυξη στη χώρα σας αυτή τη στιγμή. Και δεύτερη ερώτηση που έχει σχέση με το θέμα το οποίο ε, και η κυρία ε, Όμεν Ρόιτεν ανέφερε. Ποιοι είναι οι λόγοι, κατά τη γνώμη σας, για τους οποίους η Τουρκία είναι απρόθυμη να συνεχίσει αυτή τη διαδικασία προσέγγισης με την Αρμενία και αναμένετε θετικές εξελίξεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Κύριος Χατζηγεωργιού δύο λεπτά. Να καλωσορίσω και εγώ τον εκπρόσωπο της Αρμενίας στο κοινοβούλιο μας. Εγώ προέρχομαι από μια χώρα, αγαπητέ φίλε, που φιλοξενεί ή μάλλον έχει μεγάλη κοινότητα Αρμενίων παρακολουθούμε χρόνια τα προβλήματα της Αρμενίας όπως εξελίσσονται στην περιοχή. Θα επικεντρώσω όμως και εγώ το ενδιαφέρον μου σε ένα-δυο ζητήματα που έχουν ήδη εγερθεί ε, αλλά καλό είναι να επαναλαμβάνονται. Το ένα είναι το πρόβλημα των ε, συμφωνιών ε, με την Τουρκία που δεν έχουν προωθηθεί ούτε στο Κοινοβούλιο της Τουρκίας ούτε, στο δικό σας. Ε, πρέπει να μας δώσετε να κατανοήσουμε πού βρίσκεται η αιτία αυτού του ζητήματος. Εμένα μου δίνεται κάποτε η εντύπωση ότι από τη στιγμή της υπογραφής αυτών των συμφωνιών στην Γενέβη από εκείνη τη στιγμή υπήρχε η εντύπωση ότι η Τουρκία δεν θα τα έφερνε ενώπιον της Μεγάλης Εθνοσυνέλευσης αλλά υπήρχε και μια αίσθηση πως ούτε και η Αρμενία θα προωθούσε. Σαν να ήταν μια συμφωνία που βόλευε εκείνη την συγκεκριμένη στιγμή για κάποιους λόγους. Να μας το ξεκαθαρίσετε να το κατανοήσουμε. Το δεύτερο με τον Ακόρνο Καραπάχ. Υπάρχουν οι αιτίε στις οποίες αναφερθήκατε που προκαλούν ένα, μια στασιμότητα. Όμως θα ήθελα να δω τι, τι διέξοδο προβλέπετε. Και αν δεν προβλέπετε διέξοδο διότι η στάση του Αζερβαϊτζάν είναι αυτή σε συνεργασία με την Τουρκία κλπ. Έχετε κάτι να εισηγηθείτε, ζητάτε κάτι <clears throat> από την, ε, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, θα κλείσω με, μια, ένα μικρό σχόλιο ε, πάνω σε μια κουβέντα του κυρίου Τάνοκ που είπε ότι το κλείσιμο των σύνορων με την Τουρκία ισοδυναμεί με το να έκλειε η Ελλάδα τα σύνορά της με την Τουρκία επειδή η Τουρκία κατέχει την, την μισή Κύπρο και απλώς να σχολιάσω λέγοντας ότι ελπίζω στην αίθουσα να μην υπάρχουν πολλοί Έλληνες ευρωβουλευτές να έχουν ακούσει την εισήγηση. Δεν υπονοώ καθόλου ότι ήταν εισήγηση προς έγκριση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Γεωργίου. Ο κύριος Μιγιάν μόνο για δύο λεπτά για να κλείσει ο πρώτος γύρος των ομιλητών. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλώς ορίσατε κύριε απραγματικά θα ήθελα και εγώ να σας ρωτήσω για το ορεινό Καραμπάχ. Έγιναν ήδη πολλές ερωτήσεις. Θα αναφερθώ σε άλλο θέμα λοιπόν. Η ελευθερία των μέσων του τύπου, το media, στη χώρα σας, πώς προχωρεί. Πρόσφατα διάβασα έκθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Λέγεται ότι γίνεται ε, πρόοδος σε θέματα δημόσιας ραδιοτηλεόρασης με περσινό νόμο όπου συμπεριλαμβάνονται διάφορες προτάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης. Αλλά υπάρχει και δικαιοστάσιο μέχρι τον Ιούλιο για τις άδειε ραδιοτηλεόρασης. Ποιες είναι οι προοπτικές, ποια είναι η λύση. Δεύτερον, Τουρκία. Δεν θα επανέλθω στο διμερές, αρκετά αναφέρθηκε. Γνωρίζετε ότι τον τελευταίο χρόνο πολλοί παρατηρητές συμφωνούν ότι στην Τουρκία κυοφορείται μια νέα διαφορετική εξωτερική πολιτική. Πολλοί λέγουν ότι είναι εμπνεύσεως του κυρίου Νταβούτογλου, του νέου Υπουργού Εξωτερικών και θα ήταν κυρίως ενίσχυση της Τουρκίας ως μεγάλη περιφερειακή δύναμη και μια νέα πολιτική απέναντι στους γείτονες και τους ε, Ρώσους και το Ιράν, ε, τη Συρία μέχρι και γιατί όχι και την Αρμενία. Εσείς το έχετε διαπιστώσει αυτό, πώς γίνεται αισθητό από το ρόλο σας που έχετε και ιδιαίτερη σχέση με αυτά. Η Τουρκία περιστρέφεται περισσότερο και προσανατολίζεται προς την πρώην Οθωμανική Αυτοκρατορία και έχει απεμπολίσει την παλιά της ιδέα για ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Ευχαριστώ πολύ. Πριν δώσω το λόγο στον ε, Πρόεδρε, θα δώσω 30 δευτερόλεπτα στον κύριο Τάνο να απαντήσει στον κύριο Χατζηγεωργίου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να απαντήσω γιατί αναφέρθηκε το όνομά μου, ίσω λόγω παρανόηση, ίσω κάπου χάθηκε στην ε, διαδικασία. Είπα ότι θα ήταν εξίσου παράλογο, σαν να έκλεινε η Ελλάδα τα σύνορά τη με την Τουρκία, επειδή υπάρχει η εισβολή της Κύπρου σε αλληλεγγύη με τους ελληνοκύπριους αδερφούς λόγω της τουρκικής κατοχής στην Κύπρο. Είμαι ε, φιλέλληνας και ε, ε, φίλος των Ελλήνων. Ίσως ο Κύπριος συνάδελφος δεν κατάλαβε. Απλώς δεν συμφωνώ με το κλείσιμο των συνόρων σε αλληλεγγύη με τρίτους, ούτως ή άλλως. Ευχαριστούμε κύριε Τάνοκ. Κύριε Πρόεδρε, αν θέλετε να παραμένετε σε 10 λεπτά στην απάντησή σα, ακόμη και αν είναι 7 οι παρεμβάσει, θα πρέπει να δείξετε εδώ πόσο ακριβεί μπορεί να είστε Θα προσπαθήσω να μοδοποιήσω τις ερωτήσεις για να δώσω γενικότερες απαντήσεις. Για το πρώτο ερώτημα. Πώς θα μπορούσαμε να ξεπεράσουμε το αδιέξοδο, το τέλμα στις σχέσεις Τουρκίας-Αρμενίας. Ξέρετε όλοι ότι πέρσι στην Ζηρίχη υπεγράφησαν δύο πρωτόκολλα πρωτόκολλα που ε, με την πρωτοβουλία του Προέδρου της χώρας, ε, της Αρμενίας, αρχικά ετοιμάστηκαν, σκοπός ήταν να αναγνωριστεί και η γενοκτονία του 1915 από τους Οθωμανούς Τούρκους και έκτοτε Ούτως ή άλλως, εμείς την ε, ε, ενίσχυση των διπλωματικών μας σχέσεων με την Τουρκία δεν την βασίσαμε στην επιβολή όρων. Τα πρωτόκολλα λοιπόν αυτά υπογράφηκαν, όμως το τέλμα στις σχέσεις μας, το αδιέξοδο, το προκάλεσε η τουρκική κυβέρνηση. Δέκα μέρες μετά την υπογραφή των πρωτοκόλλων, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών έκανε δηλώσεις και είπε ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν διπλωματικές σχέσεις με την Αρμενία, ούτε θα ανοίξουν τα σύνορα, εφόσον παραμένει ανεπίλητη η διένεξη του Καραμπάχ. Αυτό ήταν το πρόσχημα της τουρκικής κυβέρνησης για την ε, πάυση της διαδικασίας. Τώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ελβετία, η Γαλλία Όλοι ήταν παρόντε στην επεξεργασία των πρωτοκόλων, όλοι παρέστησαν στην τελετή υπογραφή των πρωτοκόλων Αρμενία-Τουρκία. Δεν υπήρχε εκεί επιβολή όρων ή κάποια άλλη αιτιολόγηση για την μη, ε, παρα... Παν... Ε, για τη μη επενέναρξη των διπλωματικών σχέσεων. Ε, και μάλιστα αυτό που όλοι λογικά περίμεναν ήταν ότι θα κυρώνονταν τα πρωτόκολλα μέσα σε ευλογο διάστημα στην Συνέλευση τη κάθε χώρα. Ε, μάλιστα ο πρόεδρος της χώρας διαβεβαίωσε ότι το κοινοβούλιο όπου το μεγαλύτερο μέρος των εδρών κατέχει το κυβερνόν κόμμα ε, θα προχωρούσε στην κύρωση των πρωτοκόλων. Τώρα, γιατί δεν περιλήφθη η κύρωση των πρωτοκόλων στην ατζέντα του Αρμανικού Κοινοβουλίου, κάτι που ρώτησε ένα άλλο συνάδελφο, να πω ότι προβλεπόταν αρχικά αυτό. Περιμέναμε την απόφαση της μόνιμης επιτροπής του Αρμενικού Κοινοβουλίου. Πριν ε, ολοκληρωθεί η διαδικασία κύρωσης. Ήταν κάτι λοιπόν που αρχικά το προβλέψαμε στην ημερήσια διαταξή μα. όμως ο πρόεδρος τη χώρα άσκησε τα, θεσμικά του, τα συνταγματικά του δικαιώματα και απέσυρε από την ατζέντα μας το θέμα αυτό. Παρέμεινε βέβαια στη μελλοντική σειρά προτεραιοτήτων μα το όλο θέμα. Η πραγματικότητα όμω είναι η εξή. Εμεί δεν έχουμε κάνει τίποτα για να παρεμποδίσουμε τη διαδικασία. Το γνωρίζετε αυτό. Δεν μπορεί να σχετίζεται το ένα θέμα με, το άλλο, με την γενοκτονία των Αρμενίων δηλαδή. Και δεν μπορεί αυτό το θέμα επίση να συνδέεται με τον Αγκόρνο Καραμπάχ. Τώρα στον κύριο Κυρίλοφ να πω ότι εμεί προσέχουμε πάρα πολύ τη διατύπωση που χρησιμοποιούμε στι δηλώσεις μας. Προσπαθούμε να ενισχύσουμε και να σταθεροποιήσουμε την ε, χώρα. Προσπαθούμε να εξεύρουμε τη σωστή ισορροπία μεταξύ ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σεβασμού του και κοινωνικών υποχρεώσεων. Δεν το πετυχαίνουμε πάντοτε, ιδίω γιατί δεν έχουμε ίσω και την ε, παράδοση, τι παραδοσιακέ πρακτικέ για κάτι τέτοιο. Συχνά το κράτος επιβάλλει περιορισμού στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για να προσπίσει τα ένομα συμφέροντά του. Όμως, κάποιες φορές επίσης, τα μέσα μαζικής, μαζικής ενημέρωσης ε, επιβάλλουν πλήγματα και στο κράτος και στο κύρος του. Αυτά είναι φαινόμενα ανεπιθύμητα και αρνητικά αλλά είναι κάτι το αναπόφευκτο σε μια περίοδο μεταβατική. Πάντως, η έκθεση για τη στρατηγική στο Νότιο Κάφκασο ήταν ένα έγγραφο που μελέτησα με ιδιαίτερη προσοχή. Και Το γεγονό ότι μίλησα για μια λανθασμένη διατύπωση στο ψήφισμα και κατηγόρησα ίσω ε, του συντάκτε του ψηφίσματο στην αρχική μου ομιλία, αυτό έχει να κάνει με τα σχόλια. Τα σχόλια που είδα για τις τρεις χώρες του Νοτιού Καυκάσου που περιλαμβάνονται στην έκθεση. Θεώρησα ότι είναι μεροληπτικά τα σχόλια αυτά. Ε, η στρατηγική, μάλλον η επίλυση του ζητήματος του Ναγκόρνο Καραμπάχ, είπαμε ότι πρέπει να είναι κάτι που το δούμε και με την αρχή εδαφικής ακεραιότητας. Αλλά δεν μπορεί αυτό να είναι πρόσχημα για να και να χρησιμοποιηθεί ως επιχείρημα στις για την επίλυση του ζητήματος. Τα κείμενα που εγκρίθηκαν το 2009 και 2010 με την ε, διαμεσολάβηση της ομάδας Μίνξ του ΑΣΕ οδήγησαν σε ένα προκαταρτικό στάδιο διαπραγματεύσεων και η αρχή της αυτοδιάθεσης αναγνωρίστηκε. Αυτό θα πρέπει να αξιοποιηθεί και στο σχεδιασμό νέας πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον Νότιο Κάφκασο. Κάτι που νομίζω ότι γίνεται μέχρι το έκθεση, κύριε Λόφ. Άλλωστε και οι διεθνεί συνθήκε και τα ψηφίσματα του ΙΑ για το κράτο δικαίου, κατά ένα λόγο, προβλέπουν. Τώρα για τι γενικέ αρχέ, τι αρχέ τη Μαδρίτη, που τις έχουμε ήδη εγκρίνει, είναι ένα σημείο αφετηρία για τις συνομιλίες μας. Ε, σοβαρά σοβαρότερες απειλές κατά της Αρμενίας πέραν των Αγκόρνο Καραμπάχ. υπάρχουν, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Αρμενία είναι εκείνη που μπορεί να εκφράσει την αλληλεγγύη της, να διαφυλάξει την ασφάλεια του λαού του Ναγκορνό Καραμπάχ. Μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια του λόγου αυτού. Από τη δική μας πλευρά των συνόρων δεν ξεκίνησε κανένα θερμό επεισόδιο. Από τη στιγμή που υπογράφτηκε η Συμφωνία Ειρήνης, το Ναγκόρνο Καραμπάχ παραμένει στα πλαίσια... Είναι, κάτι που... είναι ένα περιοχή που έχουμε σεβαστεί προς την κυρία ε, αυτή και σεβόμαστε την αρχή της εδαφικής ακεραιότητας, της αυτοδιάθεσης και της μη χρήσης βίας. Τώρα, γιατί η Τουρκία είναι απρόθυμη να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις με την Αρμενία. Τι να σας πω. Η Τουρκία υφίσταται μεγάλη πίεση από την κυβέρνηση του Αζερπαϊτζάν. και οι πολιτικές δυνάμεις αυτός δηλώνουν ότι το Αζερβαϊτζάν και η Τουρκία είναι αδελφές χώρες. Και η Τουρκία θέτει ε, τα συμφέροντα αυτά και τη συνεργασία της με το Αζερβαϊτζάν υπεράνω των υπογραφών που έχει βάλει στη Ζηρίχη. Και η Τουρκία είναι ενεχόμενο μέρος. Εμείς είμαστε διατεθειμένοι να ε, κυρώσουμε τα πρωτόκολλα ακόμα και σήμερα, αρκεί η Τουρκία να συμφωνήσει. Και πάλι, γιατί δεν μπήκαν τα πρωτόκολλα στην ημερήσια διάταξη της Αρμενικής Βουλής και εγώ διερωτώ και έκανα και αυτή την ερώτηση ο ίδιος. Αλλά συμπεριλήφθησαν και μπήκαν στην ημερησία διάταξη μέχρι που τα απέσυρε ο πρόεδρος μετά από απόφαση του συνταγματικού δικαστήρου είχαν εγγραφεί. Σε ό,τι αφορά τα μέσα ενημέρωση τώρα και το πλαίσιο στο οποίο λειτουργούν. Έχουμε ε, υποβάλει και εγκρίνει πολλές τοπολογίες στον αντίστοιχο νόμο και στην αντίστοιχη επιτροπή του Συμβουλίου της Ευρώπης, ατύπως. Και το Σεπτέμβριο θα γίνει η συζήτηση στη Βουλή βάσει των ε, Επιτροπών και του Συμβουλίου της Ευρώπης που άτυπα διαβουλευτήκαμε για να δούμε πώς θα πρέπει να αλλάξει ο εκλογικός νόμος. Και στα τέλη του φθινοπόρου θα έχουμε αποτελέσματα. Σε ό,τι αφορά τώρα για το νόμο για τη ραδιοτηλεόραση, πριν από ένα μήνα τροποποιήθηκε και μέχρι τις 20 Ιουλίου θα πρέπει να προκηρύξουμε διαγωνισμό για την αδειοδότηση ραδιοτηλεπτικών σταθμών και πάλι πιστεύουμε ότι το φθινόπωρο θα τροποποιηθεί αυτή η νομοθεσία. Ε, Τελευταία ερώτηση σχετικά με την Τουρκία και τις περιφερειακές της ε, βλέψεις. Νομίζω ότι φιλοδοξεί η Τουρκία σε αυτό, το δείχνει και προσπαθεί να είναι ε, και ενδιάμεσος διαμεσολαβητής ε, στη διένεξη του Ναγκόρνο Καραμπάχ. Για μας αυτό είναι απαράδεκτο. Αυτό το θέμα μπορεί να λυθεί μόνο με διαμεσολάβηση του ΟΑΣΕ και της ομάδας του Μίνσκ. Δεν επιθυμούμε να δούμε την Τουρκία ως τέταρτο διαμεσολαβητή στην υπόθεση αυτή του Ορνού Καραμπάχ και των ενευτικών ε, συνομιλιών. Η Τουρκία προσπαθεί να ενισχύσει τον περιφερειακό της ρόλο, αλλά δεν ε, μας βρίσκει σύμφωνο σε αυτό. Σας ευχαριστούμε. Περνάμε στο δεύτερο μέρος της συζήτησης με την παρέμβαση του κ. Γκίμπου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ε, ότι καταρχάς ευχαριστώ το εξοχό κύριο Πρέσβη για την παρουσίαση. Από το 2006 νομίζω έχετε κάνει αρκετές πρόοδους από τότε που η χώρα σας εντάχθηκε στην ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας και στο ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό μέσο. Εκπονήθηκαν εθνικά προγράμματα και προγραμματα ανατολισμου προσανατολισμού 2007-2010. Τώρα πώς έρχεστε να αξιολογήσετε την εφαρμογή, την υλοποίηση αυτών των προγραμμάτων που εντάσσονται στην Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας. Επίσης συμμετέχει και στην Ανατολική Εταιρική Σχέση Αρμενία. Και αυτό τον καιρό περιμένουμε ακόμα να τεθεί σε ισχύ ε, ε, η Euronest. Σας ερωτώ, πώς βλέπετε εκεί τη συμμετοχή της Λευκορωσίας στη Euronest πάντα. Δεδομένου ότι οι εκλογές εκεί δεν είναι δημοκρατικές και η εκπροσώπηση δεν είναι αναλογική και πλήρης, κύριε Πρόεδρε. Και ένα τελευταίο θέμα. Τι λέτε, ποια είναι η προσωπική σας άποψη για το ρόλο που θα πρέπει να διαδραματίζουν οι χώρες του Νοτιού Καυκάσου, συμπεριλαμβανομένης και της ε, ε, Αρμενίας, στη διαφοροποίηση πηγών ε, ενέργειας και οδών ενέργειας προς την Ευρώπη. Ε, να έχουμε και ένα είδος ενεργειακής ισορροπίας. Και ένα τελευταίο. Είπε ο συγητής ότι στην έκθεσή του για την Αρμενία θα ήθελε να επικεντρωθεί στο μέλλον, γιατί αυτό είναι ο καλύτερος ιονός για το πώς θα προχωρήσουμε προς το μέλλον. Αλλά δεν μπορεί κανείς να αποφύγει τελείως ορισμένα θέματα του παρελθόντος. Και θέλω να σας ρωτήσω για ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πάντα ανέκαθεν σημαντικό στοιχείο για την Ευρωπαϊκή Ένωση και με τη συνθήκη της ε, Λισαβόνας. Αυτό δεν ήταν πάντα γεγονό, έτσι, σοβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θέλω να εκφράσω τη χαρά μας που βρίσκεται εδώ παρόν εκπρόσωπος του Αρμενικού Κοινοβουλίου και του λαού της Αρμενίας. Παρακολουθούμε την πρόοδο της Αρμενίας, ιδίως στις περιοχές, ε, στους τομείς που ήδη αναφέρθηκαν ε, δικαιοσύνης, ε, οικονομίας, περιφερειακής συνεργασίας, και ακούμε ότι η Αρμενία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να επιληθούν τα προβλήματα που υπάρχουν στην περιοχή και για να βελτιώσει τη δυνατότητά της να καταλήξει σε καλύτερη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιαίτερα μετά τη Συμφωνία Σύνδεσης. Θα ήθελα να επαναλάβω ένα θέμα το οποίο ανέφεραν και άλλοι συνάδελφοι ευρωβουλευτέ σήμερα. Πριν από ένα χρόνο, εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θεωρούσαμε ότι είναι ανοιχτά τα σύνορα μεταξύ Τουρκίας και Αρμενίας, ότι θα υπήρχαν διπλωματικές σχέσεις και ανταλλαγή πρέσβεων μεταξύ των δύο χωρών και θεωρήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι πρόκειται για μια νέα πολιτική της Τουρκίας ε, για να ρυθμιστούν τα προβλήματα μεταξύ Τουρκίας και γειτονικών χωρών, βάσει αυτό που μας είχε πει και ο πρέσβης της Τουρκίας. Από αυτά που μας λέτε σήμερα, ε, βλέπουμε ότι μετά την υπογραφή των πρωτοκόλων δεν έχει υπάρξει πραγματική προσπάθεια για να καταλήξετε σε επιτυχία για αυτά τα θέματα, για να υπάρξει άνοιγμα των συνόρων και για να ε, υπάρξουν και διπλωματικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών. Πώς νομίζετε ότι μπορεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή η Ευρωπαϊκή Ένωση να βοηθήσει την Αρμενία ε, να οδηγηθεί σε επιτυχία και να βελτιώσει τις σχέσεις με την Τουρκία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Μαυρονικόλα. Ο κύριος Κόβατσεφ, δύο λεπτά. Ευχαριστώ Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε της Βουλής. Χαίρομαι πάρα πολύ που ήρθατε εδώ να μας επισκεφτείτε σήμερα. Στη χώρα μου υπάρχει μεγάλη αρμενική κοινότητα, είμαι από τη Βουλγαρία και γι' αυτό ε, δείχνουμε ιδιαίτερη ευαισθησία στα θέματα αυτά και στο τι συμβαίνει στην Αρμενία. Είναι σε πολύ δυσχερή θέση αυτή τη στιγμή η Αρμενία στην περιφέρεια γενικά, αλλά και στο εσωτερικό της χώρας έχετε δυσκολίες. Έχετε βεβαίως ε, κάνει μεγάλες προόδρους προς τον ε, εκδημοκρατισμό, την αλλαγή του εκλογικού νόμου, την καταπολέμηση της διαφθοράς σε όλο το σύστημα, ανεξαρτησία του τύπου κλπ. Η Αρμενία εργάζεται σωστά και συνεργάζεται με εμπειρογνώμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν μπορώ παρά να σας ανθαρρύνω και στο μέλλον να συνεχίσετε προς την κατεύθυνση αυτή. Διεθνώς, υπάρχει το θέμα της διένεξης του Αγκόρνο Καραπάχ. Νομίζω ότι υπάρχουν τρεις αρχές που είναι εξίσου σημαντικές και αυτές είναι η εδαφική ακαιρεότητα, η, ανεξαρτησία, η, η μάλλον, αυτοδιάθεση και η μη βία. Εύκολο δεν θα είναι ούτε ταχύ, αλλά θα πρέπει να είμαστε υπομονετικοί και με υπομονή και επιμονή να σταθούμε στις τρεις αυτές αρχές. Βεβαίως δεν μπορώ να είμαι ούτε ικανοποιημένος ούτε ευχαριστημένος να επικαλείται μια δύναμη τη περιοχής εκθέσει του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να ενισχύει τι θέσει τη, όλοι κατανοούμε τι εννοώ. Και θα ήθελα να σας ε, ρωτήσω το εξή. Δεν νομίζετε ότι θα ήταν καλύτερο για την Αρμενία να επικυρώσει τα πρωτόκολλα και παρόλα αυτά να φέρει ε, την Τουρκία σε ακόμα μεγαλύτερη διεθνή πίεση επικυρώνοντας αυτά τα πρωτόκολλα και να είναι πλέον το μπαλάκι στο γήπεδο της Τουρκίας. Και η Τουρκία διαφημίζει πλέον μια πολιτική μηδενικών διενέξεων. Όλοι την κάνει και πραγματικότητα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Κόβατσεφ. Ουγγουρεάνου παρακαλώ. Εισηγητής για τη στατική ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης Μαύρης Θάλασσας. Για δύο λεπτά. Απουσιάζει. Ο κύριος Λαντσμπέργης τότε. Για ένα λεπτό, γιατί ε, έχουμε ξεπεράσει το χρόνο μας, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν βλέπουμε πρόοδο προς την ειρήνη μεταξύ Αρμενίας και Αζερβαϊτζάν. Είναι μάλλον ψυχρός πόλεμος, παγωμένος πόλεμος και ανά πάσα στιγμή μπορεί να αποψυχθεί. Είναι ολογιακή βόμβα. Δεν θα πρέπει να το αφήνουμε αυτό έτσι να διαιωνίζεται. Γιατί δεν ξέρουμε πότε θα αποψυχθεί. Εάν ο αγωγός Ναμπούκο γίνει πραγματικότητα, τότε ε, ο καλύτερος τρόπος να σταματήσει αυτό το σχέδιο θα ήταν ένας νέος πόλεμος στο Νότιο Κάφκασα ε, ε, κατά του Αζερμπαϊτζάν και θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί η Αρμενία ως αποδιοπομπαίος τράγος σε αυτά τα νέα σχέδια ε, και τα πολεμικά παιχνίδια. Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης εκεί. Το λαμβάνετε αυτό υπόψη, το εξετάζετε στην Αρμενία μεταξύ της πολιτικής ελίτ. Πώς να μην γίνεται έτσι ένα θύμα

σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή πολιτική γειτονία. Με ρωτήσατε. Και πώς αξιολογούμε τα πρώτα έτη. Ήμουν από τους πρώτους προέδρους ε, κοινοβουλίων που ε, συμμετείχα από την αρχή σε αυτή την προσπάθεια και για τη Euronest συνεργαζόμαστε με τις αρμόδιες υπηρεσίες με τρόπο επικοδομητικό και θετικό και είμαι σε επαφή και τηλεφωνική με τον πρόεδρο Μπούζεκ για τη Euronest και για τη Λευκορωσία. Νομίζω ότι οι έξι χώρες θα πρέπει να συναντηθούν και να συζητήσουν τα διαδικαστικά προβλήματα. Εμείς κάναμε κάποιες προτάσεις τροποποίησης του σχεδίου κανονισμού της Euronest συζητήσαμε και τη συμμετοχή της Λευκορωσίας και η θέση μας είναι, επαναλαμβάνω, οι έξι ενδιαφερόμενες χώρες να συνέλθουν και να συνεννοηθούν. Για τη Λευκορωσία και τη συμμετοχή της ή άλλες επιλογές που ενδεχομένως να έχουμε, ας πούμε, πέντε εκπροσώπους κυβέρνησης και πέντε της αντιπολίτευσης, αυτό δεν έγινε δεκτό από την κυβέρνηση της Λευκορωσίας. Παρ' αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε και να εφαρμόσουμε αυτή την πρωτοβούλια. Αυτό το συμφωνήσαμε στις Βρυξέλλες. Αν χρειαστεί θα γίνει και άλλη ε, συνεδρίαση των έξι πρόεδρων και το υποβάλλω και γραπτό αυτό στον πρόεδρο Μπούζεκ. Αν χρειαστεί κάνουμε ό,τι μπορούμε για να εφαρμόσουμε τη UNORS και να την υλοποιήσουμε στην πράξη. Με ρωτήσατε πώς εκτιμώ εγώ την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα. Κοίταξε, οι απόψεις ποικίλουν. Υποτίθεται ότι έχουμε πολιτικούς κρατουμένους ή καταδίκους για τις πολιτικές του Οι πολίτες που κρατούνται ή καταδικάζονται έχουν καταδικαστεί διότι έχουν τελέσει κάποιες αξιόπινες πράξεις. Δεν έχουμε πολιτικούς κρατουμένους, ούτε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι όλοι ίσοι απέναντι στον νόμο στην Αρμενία. Εργαζόμαστε με το Συμβούλιο της Ευρώπης και τον Τόν Σαμιόρκ που είναι αρμόδιος για τα ανθρώπινα δικαιώματα και προωθούμε τις δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις, στα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου. Έχουμε άλλωστε επιδείξει πολιτική βούληση να ε, υλοποιήσουμε αυτές τις μεταρρυθμίσεις και η κυβέρνησή μας θέλει η δημοκρατία της Αρμενίας να καταστεί μέλος ε, της ευρωπαϊκής οικογένειας στο μέλλον. Για την Τουρκία τώρα και κατά πόσο δεν υπάρχει πρόοδος ή αν μπορεί να μας βοηθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση η σχέση μας με τις Τουρκίες. Με την Τουρκία, ε, Πρόοδος όχι, δεν υπάρχει, διότι η τουρκική κυβέρνηση ακολουθεί άφρονα πολιτική. Είχαμε συμφωνήσει να υπογραφούν και να ακυρωθούν τα πρωτόκολλα χωρίς κανένα πρώτερο όρο και προϋποθέσεις. Αυτή τη στιγμή που συζητούμε εδώ, εμείς είμαστε πρόθυμοι να κυρώσουμε τα πρωτόκολλα που έχει υπογράψει ο υπουργό Εξωτερικών μας. Ωστόσο, δεν βλέπω την Τουρκία να επιδεικνύει την ίδια πολιτική βούληση. Η Αρμενία είναι ανα πάσα στιγμή έτοιμη να υπογράψει και να κυρώσει. Αυτή τη στιγμή θα κυρώσει και η Τουρκία τα προλόκαλα αυτά. Και, καλούμε, και παρακαλούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να πιέσει την τουρκική κυβέρνηση να κυρώσει τα πρωτόκολλα τα οποία ήδη έχει υπογράψει και έχει δώσει και τη σύμφωνη γνώμη της χωρίς καμία προϋπόθεση. Έχει έρθει η ώρα της κύρωσης πλέον των πρωτοκόλων αυτών. Διαφωνώ με κάποιους συναδέλφους που προτείνουν να κυρώσουμε τώρα εμείς τα πρωτόκολλα και να φέρουμε σε ακόμη πιο δύσκολη θέση την Τουρκία. Όχι. Εμείς έχουμε κάνει το πρώτο βήμα. Ο πρόεδρος της Αρμενίας ε, έτεινε χείρα ε, προς την Τουρκία, προσκάλεσε την Τουρκία να συνεννοηθεί με την Αρμενία, να ε, συνάψουμε σχέσεις από το 1993 θυμάστε. Έχει κλείσει τα σύνορα η Τουρκία. Πριν από 17 και πλέον έτη. Θα πρέπει να τα γνωρίζουν όλοι εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και να συμφωνείτε ότι δεν μπορούμε τον 21ο αιώνα να έχουμε κλειστά σύνορα και θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να πιέσει την Τουρκία να ανοίξει τα σύνορα με την Αρμενία. Δεν πρόκειται εδώ για μια χώρα που ε, φιλοδοξεί να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Περί αυτού δεν, συζητάμε. Μια χώρα που είναι υποψήφια να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση κρατάει κλειστά τα σύνορά της με μια ε, χώρα της. Και ως πρόεδρος ε, της Αρμενικής Βουλής εγώ είμαι αντίθετος με την κύρωση από πλευρά Αρμενία των πρωτοκόλων, γιατί είμαστε πεπισμένοι ότι ακόμα και αν τα κυρώσουμε, η τουρκική κυβέρνηση δεν πρόκειται να το πράξει. Και θα προσπαθήσουν να καταχραστούν τις κατάστασης αυτής και των πρωτοκόλων για να ορίσουν τον εαυτό τους διαμεσολαβητή στο Ναγκόρνο Καραμπάχ μεταξύ Αρμενίας και Αζερβαϊτζάν. Ε, για μας είναι απαράδεκτο, σας είπα αυτό. Δεν μπορούμε να δούμε την Τουρκία ως διαμεσολαβητή στην διάνοιξη αυτή. Και ένα τελευταίο για τη διάνοιξη στο Ορεινό Καραμπάχ και κατά πόσο μπορούν να επαναληφθούν εκεί οι εχθροπραξίες. Όπως είπα και στην πρωτομιλία μου και το επαναλαμβάνω, ο πρόεδρος του Αζερβαϊτζάν, ο κύριος Αλίεφ και άλλοι αζέρι πολιτικοί δεν χάνουν ευκαιρία να κάνουν αιμοδιψείς και πολεμοχαρείς ε, δηλώσεις και προσπαθούν να μας προκαλέσουν. Τώρα που συζητούμε εδώ είναι πιθανό να πυροβολούν στα σύνορα ελεύθεροι σκοπευτές και χρησιμοποιούν τα έσοδα από το πετρέλαιο στο Αζερβαϊτζάν για να στήσουν στρατό. Και δεν βλέπω αντίστοιχη επικριτική αντιμετώπιση ή απόκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή διεθνείς οργανισμούς. Δεν βλέπω να καλεί κανείς το, το να σταματήσει τις προκλήσεις και ε, τις πολεμοχαρείς δηλώσεις. Και πάλι πιστεύω ότι τον 21ο αιώνα η πόλεμη δεν είναι λύση για κανένα πρόβλημα. Ακόμα υφιστάμεθα τις συνέπειες του πολέμου 91-94 που ξεκίνησαν ε, οι αρχές του Αζερβαϊτζάν. Και καλώ τους συναδέλφους να το σκεφτούν αυτό. Να αποκλειστεί οποιαδήποτε χρήση βίας. Δεν είναι λύση η βία. Θα πρέπει να το πούμε αυτό και στην κυβέρνηση του Αζερβαϊτζάν. Οι νευτικές συνομιλίες είναι ο δρόμος προς τη λύση. Εμείς θέλουμε ειρήνη με τους γειτονές μας. να λύσουμε όλα τα ζητήματα με τις ειρηνευτικές συνομιλίες. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε, Πρόεδρε. Η συνάντηση αυτή ήταν ιδιαίτερα επικοδομητική, διεξοδική, ενημερωτική. Θα έχουμε όμως και άλλες συναντήσεις στο μέλλον για να εμβαθύνουμε τη σχέση συνεργασία μας. Ειλικρινής ευχές από πλευράς μας για την τελευταία σας ε, δήλωση για τη διαδικασία ειρήνευσης στην περιοχή. Ελπίζουμε όλες οι κρεμούσες γυναίξεις να επιληθούν σύντομα και εμείς να μπορέσουμε να συνεισφέρουμε ω Ένωση προς την σωστή κατεύθυνση. Σας ευχαριστούμε λοιπόν όλους ε, για τις παρεμβάσει σα και αφήνω το λόγο στον κύριο Πάσκου για την συνέχεια της μερικής διατάξης. Thank you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 Uh, uh, Θα ήθελα να καλωσορίσω την εξοχότητά του τον πρέσβη Μοχάμετ Τζαουάντ Αλντορεκή, πρέσβη του Ιράκ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όπως γνωρίζετε, ε, η κατάσταση Χρειάζεται κάποιες επεξηγήσεις. Οι εκλογές έχουν γίνει εδώ και κάποιους μήνες και δεν έχουμε ακόμη τελικά αποτελέσματα. Επομένως και προς εμάς αλλά και προς όλους θα ήταν ε, καλό να έχουμε κάποιες εξηγήσεις. Και σήμερα είναι η τελευταία προθεσμία για την εκλογή του Προέδρου εφόσον βέβαια είχαν ανακοινωθεί προηγουμένω τα αποτελέσματα. Θα ήθελα να ζητήσω από, τον, από την εξοχότητα του τον κύριο Πρέσβη να ασχοληθεί με τα θέματα αυτά στην παρέμβασή του και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η συζήτηση. Και υπενθυμίζω στους συναδέλφους ότι έχουμε στη μερίσια διάταξη άλλο ένα σημείο. Για να μην καθυστερήσουμε το λέω αυτό. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, Αγαπητοί κύριοι και κυρίες Ευρωβουλευτές, κυρίες και κύριοι, καταρχήν θα ήθελα να με επιτρέψετε να ευχαριστήσω τον πρόεδρο Αλμπερτίνη που μου δίνει αυτή την πολύτιμη ευκαιρία να απευθύνω το λόγο στα μέλη της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων για την κατάσταση όπως αναπτύσσεται στη χώρα μου και για τις δεμερείς σχέσεις μεταξύ του Ιράκ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πραγματική χαρά για μένα που λαμβάνω το λόγο ενώπιόν σας. Μετά από 35 χρόνια βίαιης δικτατορίας και αυταρχικού καθεστώτος, κατά την οποία το Ιράκ απομονώθηκε από τον υπόλοιπο πολιτισμένο κόσμο και κατά τα οποία ταχαίως επιδεινώθηκαν το επίπεδο διαβίωσης, η εκπαίδευση, η υγεία και άλλοι ζωτικοί τομείς, το Ιράκ άρχισε να αναπνέει τον αέρα της ελευθερίας και της δημοκρατίας, αλλά σε ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον, καθώς ε, ακολούθησε ένα κύμα χωρίς προηγούμενο βάρβαρης τρομοκρατίας που έπνιξε τη χώρα από, με προέλευση από διάφορα μέρη του κόσμου μέσω των γειτονικών μας χωρών με υποστήριξη και χρηματοδότηση από πολλές πηγές. Και μετά από ακόμη 7 δύσκολα χρόνια κατά τα οποία πολλά συνέβησαν και κάποια στιγμή φάνηκε να σταματάει ο χρόνος όταν τρομοκράτες και ένοπλες παραστατιωτικές οργανώσεις επικρατούσαν σε πολλούς ε, τομείς, σε πολλές περιοχές της Βαγδάτης και σε άλλες μεγάλες πόλεις εκατοντάδες Ιρακινών σκοτώθηκαν και εκατοντάδες ε, εγκατέλειπαν καθημερινά τη χώρα. Οι Αλ-Κάιντα και οι σκληροπυρηνικοί ανταμιστές έκαναν ε, ό,τι μπορούσαν για να δημιουργήσουν τις συνθήκες για μια διένεξη που θα δίχαζε και δημιουργούσαν το σκηνικό για ένα εμφύλιο πόλεμο. Και πολλοί θεωρούσαν το Ιράκ φαύλο κράτο. Τελικά δεν συνέβη αυτό και η τρομοκρατία άρχισε να χάνει έδαφο ε, καθώ άλλαζαν τα πράγματα. Ήταν ένα πραγματικό θαύμα, όπω είπε ο πρόεδρο τη Γαλλία. και αφού δεν επήλθε εμφύλιο πόλεμο στο παρελθόν, δεν πρόκειται ποτέ στο μέλλον να επέλθει εμφύλιο πόλεμο. Έχει βελτιωθεί η κατάσταση από πλευρά ασφαλεία. Η Αλκαίδα και οι περιστατιωτικέ δυνάμει έχουν λάβει ισχυρά πλήγματα και παρότι έχουν αποδυναμωθεί, συνεχίζουν να είναι επιζήμιε οι δραστηριότητέ του και ακόμη μπορούν να περνάνε τα σύνορα από γειτονικέ χώρε. Από ό,τι ακούσαμε κατά τέλη του 2011 η ημερομηνία απόσυση όλων των ξένων στρατευμάτων από το Ιράκ σύμφωνα με τη συμφωνία Σόφα που υπεγράφει μετά από έντονε διαπραγματεύσει μεταξύ των κυβερνήσεων του Ιράκ και των Ηνωμένων Πολιτειών. Και είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι η ασφάλεια, οι υπηρεσίε ασφαλεία στο Ιράκ και οι ένοπλε δυνάμει ε, έχουν καλή κατάρτιση, ε, καλή προετοιμασία και έχουν αναλάβει τι ευθύνε, τι αρμοδιότητε από τι δυνάμει των Ηνωμένων Πολιτειών και εργάζονται σχεδόν ανεξάρτητα πλέον. Το Ιράκ, κυρίε και κύριοι, έχει κάνει τα πρώτα του βήματα στο δρόμο τη δημοκρατία και είναι αποφασισμένο να συνεχίσει παρά το υψηλό κόστο, όχι μόνο με την καταπολέμηση τη τρομοκρατία για λογαριασμό του ελεύθερου κόσμου, αλλά και χάρη στη συνεχή ξένη παρέμβαση στι εσωτερικέ του υποθέσει και ιδίω από γειτονικέ χώρε. Όχι μόνο διότι πολλοί στην περιφέρεια δεν χαιρετίζουν τη δημοκρατία στο Ιράκ, αλλά ε, και διότι επιθυμούν να βάλουν πόδι στη χώρα και να διαμορφώσουν το μελλοντικό Ιράκ σύμφωνα με τα δικά του συμφέροντα. Μετά από 8 χρόνια ανόητου πολέμου με το Ιράν και την εισβολή στο Κουβέιτ, οι υποδομέ ε, σχεδόν καταστράφηκαν πλήρως. Το νέο Ιράκ είναι αποφασισμένο να έχει καλέ σχέσεις με όλους τους γείτονε επί τη βάση του αμοιβαίου σεβασμού, των αμοιβαίων ε, συμφερόντων και τη μη παρεμβολή στις εσωτερικέ υποθέσει άλλων χωρών. Πιστεύουμε ότι πρέπει να προωθήσουμε αυτή την πολιτική, γιατί αυτό θα εξυπηρετήσει τα συμφέροντα όλων των ενδιαφερομένων χωρών και θα διασφαλίσει τη σταθερότητα σε μια περιφέρεια που είναι σημαντική για τον υπόλοιπο κόσμο, εφόσον είναι η περιοχή που παρέχει μεγάλο ποσοστό του ενεργειακού τους πλούτου των ενεργειακών τους αναγκών αυτή η μεταβατική διαδικασία είναι δύσκολη και πολλέ προκλήσεις συνεχίζουν να υπάρχουν για τη χώρα μας. Το νέο κοινοβούλιο και η κυβέρνηση θα πρέπει να αντιμετωπίσουν αυτές τις προκλήσεις, όπως είναι το να παλέψουν για την καλή διακυβέρνηση, να διαφοροποιήσουν τις πηγές πλούτου και να μην εξαρτώμεθα μόνο από το πετρέλαιο σαν έσοδο για τη χώρα μα, να δώσουν στη χώρα καλύτερε υπηρεσίε και να βελτιώσουν το επίπεδο ζωή. και Υπάρχουν παράλληλα πολλά πολιτικά διέξοδα όπως ε, το ευαίσθητο και πολύπλοκο θέμα του Κυρκούκ, επίμεχες περιοχές, καθώς και θέματα όπως τροποποίηση του συντάγματος, ενεργειακή νομοθεσία κλπ. Πολλές ε, βασικές, νομοθεσίες, συμφωνίες έχουν υπογραφεί με μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείε για να αυξηθεί η παραγωγή πετρελαίου και παρόμοιε συμφωνίες για την εκμετάλλευση του πλούτου σε φυσικό αέριο θα υπογραφούν σύντομα. Κυρίε και κύριοι, το Ιράκ είναι πολύπλοκη χώρα. Είναι μια χώρα με πολλέ εθνότητε, πολλέ πατρίε, θρησκείες και πολλές γλώσσες, όπως ήταν επί χιλιάδες χρόνια. Το ευρύ αυτό φάσμα θα έπρεπε να είναι μια πηγή πλούτου και διαφορετικότητας, εάν το προσεγγίσουμε από, το σωστό, από τη σωστή οπτική γωνία, με την αποδοχή και σεβασμό των πιστεύω και των δικαιωμάτων των υπολείπων. Οι πολίτες του Ιράκ και ιδίως οι πολιτικοί θα πρέπει να έχουν αμοιβαία εμπιστοσύνη και να καταφύγουν σε διάλογο και σε συμβιβαστικές λύσεις. Η διαδικασία της Εθνικής Συμφιλίωσης και Ενότητας είχε ξεκινήσει και θα έπρεπε να αντικατοπτρίζεται στο σχηματισμό της νέας κυβέρνησης που θα, έπρεπε, θα πρέπει να είναι πολυσυλλεκτική και αντιπροσωπευτική όλων των διαφορετικών συνιστοσών του λαού του Ιράκ. Οι σχέσεις μεταξύ Ιράκ και Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, εξελίσσονται με τρόπο ικανοποιητικό. Οι διαπραγματεύσει ε, για την Συμφωνία Εταιρική Σχέση και Συνεργασία ολοκληρώθηκαν πριν από λίγο καιρό και ελπίζουμε ότι θα μονογραφεί και θα υπογραφεί σύντομα αυτή η συμφωνία. Η συμφωνία αυτή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο των διαμερών μας σχέσεων και θα ήθελα να υποφεληθώ τις ευκαιρίες για να ευχαριστήσω όλους τους εμπειρογνώμονες της Επιτροπής, του Συμβουλίου και των Προεδριών που δούλεψαν σκληρά με τους Ιρακινούς ομολόγους για να επιτύχουν αυτό το στόχο. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω το προσωπικό της EU Just Lex για την θεμελιώδη συμμετοχή τους στο να παγιώσουν το κράτος δικαίου στη χώρα μου. Ένα μνημόνιο συνεργασία για την ενέργεια υπεγράφει μεταξύ του Ιρακινού Υπουργείου Πετρελαίου και τη Επιτροπή Ενέργεια και ελπίζουμε ότι θα ανοίξει το δρόμο για μελλοντική συνεργασία σε αυτό το σημαντικό τομέα. Ενώ το Ιράκ, κυρίε και κύριοι, κοιτάζει προ το μέλλον και προσβλέπει σε μια ειδική σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση από όλε τι απόψει, ε, χαιρετίζει την ε, υποστήριξη τη Ευρωπαϊκή Ένωση ε, να βοηθήσει τη χώρα να αποκτήσει πλήρη κυριαρχία, απελευθερώνοντάς το από το άχθος του κεφαλαίου 7 της Χάρτας των Ηνωμένων Εθνών που επευλήθη στο Ιράκ κατά το προηγούμενο καθεστώς και προσβλέπει σε ευρωπαϊκές επενδύσεις και συμμετοχή στη διαδικασία ενοικοδόμησης μιας χώρας που έχει όλο το δυναμικό και ανθρώπινους και φυσικούς πόρους να γίνει σύγχρονο δημοκρατικό κράτος. Κυρίε και κύριοι, θα ήθελα τώρα να θίξω ένα σημαντικό θέμα για τις διμερείς σχέσεις, για τις σχέσεις μεταξύ του ε, Ιρακινού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που τα τελευταία χρόνια έχουν εξελιχθεί με, εξελιχθεί με ταχύς ρυθμούς και με μεγάλη ε, χαρά και ευχαρίστηση θέλω να επενέσω ε, τις προσπάθειες του Προέδρου και των μελών της προηγούμενης αντιπροσωπείας για τις σχέσεις με το Ιράκ που βοήθησαν να προσεγγίσουν αυτοί οι δύο δημοκρατικοί θεσμοί δίνοντα ευκαιρίε σε βουλευτέ από το Ιράκ να υποφεληθούν από την πλούσια εμπειρία των διαφόρων επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Μέσω της διοργάνωσης πολλών επισκέψεων ε, κοινοβουλευτικών ε, αντιπροσωπιών από το Ιράκ και επιδεικνύοντας ηθική υποστήριξη της πολλές τους επισκέψεις ε, στη Βαγδάτη. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω την Βαρόνι Νίκολσον, την Άννα Γκόμες, τον Νικολάη Μιλάτνοφ και άλλα μέλη της προηγούμενης αντιπροσωπείας. Και εδώ ελπίζω ότι δεν θα προσβάλλω κανένα μέλος του Κοινοβουλίου, εκφράζοντας την ειλικρινή μου ευχή, που είναι επιθυμία και πολλών μελών της αντιπροσωπείας, η τωρινή προεδρία της αντιπροσωπείας για τη σχέση με το Ιράκ να συνεχίσει την αποστολή που έχει αναλάβει και να ζητήσουμε από τον πρόεδρο να μην μεροληπτεί, να μην προωθεί τις απόψεις και τα συμφέροντα κάποιας πολιτικής οντότητας στο Ιράκ και να τηρεί ίσες αποστάσεις από τις διαφορετικές Ιρακινές πολιτικές ε, οντότητες και να μην ε, προσβάλλει το λαϊκό αίσθημα στο Ιράκ και ε, καθώς και ε, τις απόψεις των εκπροσώπων των πολιτών στο Κοινοβούλιο του Ιράκ, συνεχίζοντας ε, να ε, παίρνει σε πολλές περιστάσεις το μέρος κάποιες οργάνωσης που θεωρείται τρομοκρατική από το Σύνταγμα του Ιράκ και που συμμετέσχε με τις αποτρόπες δυνάμεις ασφαλείας του προηγούμενου καθεστώτος στη δίαιη και ανηλεή καταστολή της λαϊκής εξέγερσης του 1991. Αυτό αποτελεί παρέμβαση στην εσωτερική πολιτική του Ιράκ και δεν θα βοηθήσει τις προσπάθειες να επιτύχουμε τη συμφιλίωση, ούτε θα βελτιώσει τις σχέσεις μεταξύ Ιράκ και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκτιμώ ιδιαίτερω, κυρίε και κύριοι, αξιότιμοι κύριοι βουλευτέ, ε, μέλη τη Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, το ενδιαφέρον σα για την κατάσταση όπω εξελίσσεται στη χώρα μου και ελπίζω ότι ε, με αξιοπιστία και με υπευθυνότητα θα συνεχίσετε να διασφαλίσετε τις διμερείς μας σχέσεις και ιδίως τις ε, υγιείς σχέσεις μεταξύ των δύο κοινοβουλίων όπως έχουν εξελιχθεί μέχρι τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Θα σας ευχαριστώ όλοι ο Πρόεδρος και θα ήθελα να αναζητήσω τώρα από τον κύριο Μάουρο που είναι ο εισηγητής για το Ιράκ να λάβει το λόγο. Έχετε το λόγο κύριε Μάουρο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον εξοχότατο κύριο Πρέσβη για την εισαγωγή του. Πρέπει να σας πω ότι Διακόπτει ο μιλητής. Φαντάζομαι ότι τώρα με ακούτε, κύριε Πρέσβη. Οπότε μπορώ να ξεκινήσω με τις ερωτήσεις μου. Και ξεκινώ από αυτό που περισσότερα από όλα μας ανησυχεί. Έχετε περισσότερες πληροφορίες εσείς από τη δική σας πλευρά για την κυβέρνηση είναι απλή ερώτηση. Θεωρείτε ότι αυτός ο σχηματισμός κυβέρνησης θα μπορούσε να επέλθει σύντομα, ως το δυνατόν συντομότερα και σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές του 2005 συγκεκριμένα θα μπορούσατε να μας δώσετε περισσότερες λεπτομέρειες σε σχέση με το τι παρεμποδίζει το σχηματισμό νέας κυβέρνησης τις συγκρούσεις, τις διαφωνίες μεταξύ του κ. Μαλίκη και του κ. Αλάουι των κομμάτων των συνιστοσών της κοινωνίας των πολιτών στο Ιράκ. Τι εμποδίζει να φτάσουμε σε ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα σύντομα και δεδομένων και των προσπαθειών που καταβάλλονται. Έπειτα, είχα μια ερώτηση σε σχέση με, την ε, νέα, με το νέο κύμα βίας παρά την ανασυγκρότηση των ε, δυνάμεων ασφάλειας. Εσεί είπατε ότι ήταν επιτυχής βεβαίω, αλλά ποια θα είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που θα έχουν να αντιμετωπίσουν από την άποψη τη ασφάλεια και εφόσον αποσυρθούν τα αμερικανικά στρατεύματα. Ήδη προετοιμάζεται αυτό. Όταν θα έχει ολοκληρωθεί, τι θα γίνει. Και έπειτα για τι μειονότητες. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα εκατομμύριο Ιρακινών που ζουν σε εκτός χώρας, στη Συρία και την Ιορδανία. Τι μέτρα θα λάβει η κυβέρνησή σα, ώστε να ενθαρρύνει τους ε, μετανάστε, τους πρόσφυγες να επιστρέψουν στη χώρα. Επαγγελματικά κίνητρα, ε, γιατί η επιστροφή των μεταναστών θα μπορέσει να βοηθήσει ενδεχομένω τη χώρα στην ανάκαμψή τη. Και σε σχέση με την προηγούμενη κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Εσεί πώ βλέπετε τι δυσκολίε που συναντήσαμε ω τώρα στι διαπραγματεύσει. και τι θεωρείτε ότι ήταν ε, σημαντικό προ προς την συμφωνία που βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση και ελπίζουμε να περατωθεί σύντομα. Βάσει των δικών σα κανόνων πρέπει να εγκρίνει το Κοινοβούλιο την υπογραφή τη συμφωνία. Ελπίζουμε λοιπόν στην Επιτροπή μα να δεχτούμε ω επισκέπτε και μέλη του Ιρακινού Κοινοβουλίου για να έχουμε μια πραγματική ανταλλαγή απόψεων μεταξύ βουλευτών από το Ιράκ και βουλευτών από το Ευρωκοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Μάουρο. Και η κυρία Γκόμες τώρα. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ και τον Πρέσβη για την πολύ ειλικρινή παρουσίαση αυτή. Μας είπε ότι το Ιράκ είναι μια χώρα πολύπλοκη. Αλλά τα πράγματα κινούνται. Στόχος είναι να μην φτάσει η χώρα πάλι στο χείλος των όσων πρόκειται να συμβούν πριν μερικά χρόνια του φαύλου κράτου. Και επίσης για τι εχθρότητες μεταξύ των φατριών που έχουμε γνωρίσει ω τώρα στο Ιράκ. Υπάρχουν ήδη διαπραγματεύσει από τι εκλογέ και μετά. Αυτό δείχνει ότι οι Ιρακινοί έχουν μάθει κάποια πράγματα από το παρελθόν. Μπορούν να επιλύσουν κάποιε δυσκολίε χωρί να επιστρέφουν ε, στι εχθροπραξίε. Η βία στο Ιράκ είναι βία κατά του Ιρακινού λαού από τρομοκρατικές ομάδες που δεν καταφέρατε να κρυζώσετε και μπόρεσαν να δρουν και μετά την εισβολή. Τώρα, η παρέμβαση έξωθεν στη χώρα σας από άλλες χώρες στο Κοινοβούλιο, στο Ευρωκοινοβούλιο, πολλοί ανησυχούν από τις παρεμβάσεις ε, από το Ιράν, αλλά κάποιοι δεν δίνουν καμία σημασία στην παρέμβαση άλλων χωρών, όπως της Σαουδικής Αραβίας ή της Συρίας ή της Τουρκίας, που πολλές φορές κάνει εφόδους στο βορρά της χώρας, ε, με αφορμή το ΠΚΚ. Ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω κατά πόσον αισθάνεστε ότι επιτελείται πρόοδος όχι μόνο για το θέμα των μεταναστών, των προσφύγων όπως σας ρώτησε ο κύριος Μάουρο, των Ιρακινών που έχουν ε, φύγει από τη χώρα, αλλά την ε, περίπτωση των εσωτερικών μετατοπισμένων. Ένα θέμα ευρύτερο από αυτό των προσφύγων. Γνωρίζω ότι αυτό έχει να κάνει και με την κατάσταση ασφαλείας. Πολλοί δεν μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους γιατί δεν αισθάνονται ακόμη ασφαλείς στον τόπο προελευσής τους. Χθες μόλις σε μια συνάντηση της αντιπροσωπείας μας για το Ιράκ με πολύ θλίψη ακούσαμε ότι μη κυβερνητικέ οργανώσεις που έχουν εργαστεί για το θέμα των δικαιωμάτων των μειονοτήτων και είχαν ελπίδες ότι παρά τις ανεξελίξεις διαπραγματεύσεις θα μπορούσαν να συνεργαστούν με Ιρακινούς βουλευτές για τα θέματα αυτά τους ερχόμενους μήνες τελικά δεν. Τελικά θα μπορέσουν να συνεχίσουν το έργο τους. Και για το μνημόνιο συνεννόησες για την ενέργεια που υπογράφηκε από την Επιτροπή. Πώς θα συνδεθεί με τις πετροπολογίες της περιοχής της ΑΚΑ. Και Εάν μπορούσατε να μας δώσετε περισσότερες πληροφορίες, τι γίνεται στις συνομιλίε σας με την κουρδική κυβέρνηση. Η επίσκεψη του πρόεδρου Μπαζάνη πρόσφατα στη Γαλλία και τη Γερμανία. Εμένα τουλάχιστον μου έδωσε ιδιαίτερη χαρά. Πιστεύω ότι αυτό είναι ένα στοιχείο που θα μπορούσε να καθησυχάσει την ε, προηγούμενη καθυποψία της Επιτροπής προς το Κουρδιστάν. Υπάρχουν πολλές ευκαιρίες εδώ. Θα μπορούσαμε να τις διερευνήσουμε για να δούμε πώς θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε τις σχέσεις όχι μόνο με την ε, περιοχή του Κουρδιστάν αλλά με το σύνολο του Ιράκ. Και περισσότερη συμμετοχή από το Κουρδιστάν και προσέλευση εμπειρογνωμόνων από το Ιράκ για να δούμε πώς μπορεί να βελτιωθεί το επίπεδο ασφαλείας εκεί. Και τέλος, να πω ότι καταλαβαίνω πολύ καλά τα όσα λέτε. Έχω κατανόηση για τα παραπονά σας ε, σε σχέση με την αντιπροσωπεία του Ιράκ, αλλά χαίρομαι ιδιαίτερα που λάβατε πρόσφατα την επιστολή μας που λέει ότι θα πρέπει κάποια κύρωση να επιβληθεί στο Ιράκ εφόσον δεν έχει βρεθεί ακόμη, δεν έχει επιληθεί το θέμα της κυβέρνησης. Αυτό όμως δεν εκπροσωπεί την ε, πλειοψηφία των μελών της αντιπροσωπείας του Ιράκ. Δεν ε, συζητήσαμε όλοι για το θέμα αυτό και χθε την αντιπροσωπεία για το Ιράκ ε, συμφωνήσαμε να προβλεφθεί διαδικασία που να μην επιτρέψει την επανάληψη των γεγονότων. Σα διαβεβαιώνω ότι εκπροσωπείται εδώ η άποψη μόνο του Πρόεδρου τη Αντιπροσωπεία και όχι τη πλειοψηφία ούτε των κυβερνήσεων που συμμετέχουν, των μελών που συμμετέχουν στην αντιπροσωπεία αυτή. Νομίζω λοιπόν ότι ήταν άδικη αυτή η κρίση τη επιστολή και παραβλέπει τις πρόοδε που έχουν επιτελεστεί παρά τις πολλαπλέ δυσκολίε που έχει συναντήσει το Ιράκ. Ευχαριστούμε. Η κυρία λοχμπιλερ πρόεδρος τη αντιπροσωπεύει για τι σχέσεις με το Ιράν. Και μετά θα διαιρέσουμε το χρόνο με τον αριθμό των αγορητών και θα σας δώσουμε και την ευκαιρία να απαντήσετε. Θα συνεχίσουμε λοιπόν με τους τέσσερις τελευταίους αγορητές. Η κυρία Λοχμπίλερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε κύριε Πρέσβη για την παρουσίασή σας. Έχω κάποιες ερωτήσεις ε, για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράκ. Στο Ιράκ ε, έχετε ένα πολύ φιλελεύθερο νόμο για την ελευθερία του τύπου. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν ε, πολλοί δημοσιογράφοι ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης ε, που αντιμετωπίζουν πολλές ποινικέ διαδικασίες που έχουν πολιτικά κίνητρα. Ε, υπάρχουν εκθέσεις ε, για επιθέσεις κατά δημοσιογράφων από άτομα με πολιτικά και αυτές οι επιθέσεις ε, ίσως είναι οργανωμένες από τις μυστικές υπηρεσίες. Αυτές είναι οι φήμες και θα ήθελα να ακούσω πώς εσείς αξιολογείτε την κατάσταση. Επίσης υπάρχουν περιπτώσεις εξοδικαστικών εκτελέσεων και, και βασανιστήριων και θα πρέπει οι υπεύθυνοι να οδηγηθούν ενώπιον του δικαστηρίου. Ε, τρίτον, ε, ε, λέγεται ότι και από το Ιράν και από την Τουρκία υπάρχουν ε, ε, επιθέσεις στο βόρειο τμήμα του Ιράκ, στην περιοχή των συνόρων του Ιράκ και ο Πρωθυπουργός Αλ Μαλίκη τον Ιούνιο είχε αναφέρει επισήμως κάτι τέτοιο και αυτές οι επιθέσεις σύμφωνα με αναφορές ε, μη κυβερνητικών οργανώσεων για τα δικαιώματα του ανθρώπου, των ανθρώπων αφορούν πολλούς αμάχους και πολλές οι οικογένειες ε, εκδιώχθηκαν από αυτή την περιοχή ακριβώς λόγω αυτών των ε, επιθέσεων. Πώς αξιολογείται την κατάσταση και η Ιρακινή κυβέρνηση τι προθέσεις έχει επί του θέματος. Και ένα τελευταίο σημείο τώρα για την κατάσταση στο Ασράφ, ε, στο Ιράκ αυτό, ε, σε αυτό το στρατόπεδο υπήρξαν δύο επιθέσεις από ό,τι έχουμε ακούσει και πολλές φορές το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει αναφερθεί και τώρα το πρακτορείο Reuters στις 11 Ιουλίου αναφέρει ότι ένα Ιρακινό δικαστήριο διέταξε τη σύλληψη 39 Μουτζαχεντίν με κατηγορίες ε, εγκλημάτων ε, κατά της ανθρωπότητας. Ε, θα ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Πρέσβη, ποιες είναι οι κατηγορίες που προσθέτονται σε αυτούς τους συλληφθέντες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Έχετε το λόγο, κύριε Πρέσβη. Και έχουμε και άλλους τέσσερις ομιλητές που θα λάβουν το λόγο στη συνέχεια. Σας ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, για τις ερωτήσεις σας. Κύριε Μάουρο, θα αρχίσω από εσάς από την τελευταία σας ερώτηση που ήταν για τις διαπραγματεύσεις. Νομίζω ότι είναι εδώ η κυρία Πατρίσια Λόμπαρτ από πλευράς ευρωπαϊκής Ευρωπαϊκή Νομίζω ότι οι διαπραγματεύσεις γίνονται πολύ καλά. Επί μία διετία με πολλούς γύρους διαπραγματεύσεων και στις Βρυξέλλες και στη Βαγδάτη. Δεν νομίζω ότι είναι μεγάλα τα προβλήματα και δυσκολίες. Ε, από τη δική μου εμπειρία πρέπει να σας πω ότι έχουμε αντίστοιχες διαπραγματεύσεις με αραβικές χώρες και άλλες χώρες στην περιοχή. Πάντα αναφέρονται προβλήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων κτλ. Στη δική μας περίπτωση δεν αναφέρθηκε κανένα τέτοιο πρόβλημα. Κάποιες λεπτομέρειες ίσονος σημασίας και ε, νομίζω ότι θα καταλήξουμε και είναι θέμα χρόνου η μονογραφή και ε, ε, η ε, ακόλουθη μακρά διαδικασία ψηφοφορία στα διάφορα εθνικά κοινοβούλια και ελπίζω και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι πάρα πολύ σημαντική η συμφωνία. Αυτή θα είναι ακρογωνιαίος λήθος των μελλοντικών μας σχέσεων και το θεσμικό πλαίσιο που θα τις διέπει. Επίσης, ερώτηση κάνατε κύριε Μάωρο για το ρόλο των ενόπλων δυνάμεων στο περασμένο καθεστώς είχαμε ένα εκατομμύριο ε, ένοπλες δυνάμεις. Γνωρίζετε ότι στη δεκαετία του 80 είχαμε πόλεμο με το Ιράν, στη συνέχεια με το Κουβέιτ, στη συνέχεια πολέμους είχαμε. ένοπλες δυνάμεις επίσης εξαπέλυαν ε, επιθέσεις προς τον ίδιο το λαό του Ιράκ και στο Νότο και στο Κουρδιστάν. Και στη συνέχεια όμως διαλύθηκε ο στρατός ε, στην αρχή της κατοχής. Και σιγά σιγά ε, καταλάβαμε ότι έπρεπε να ανασχηματίσουμε στρατό, γιατί και οι Αμερικανοί δεν ήθελαν να μείνουν ε, εκεί για περισσότερο διάστημα από όσο χρειάζεται. Πριν από ένα ε, έτος και πλέον είχαμε πολύ δύσκολες διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τελικά ε, καταλήξαμε σε μια συμφωνία πάρα πολύ ιδιαίτερη. Και είπε ο Αμερικανός πρέσβης ότι μας αφεμάξατε, γιατί ήταν πάρα πολύ σκληρή τελικά η συμφωνία και σε σχέση ε, τύπου συμφωνιών με την Ιαπωνία και την Νότια Κορέα έχουν κάνει ε, τέτοιες συμφωνίες οι Ηνωμένε Πολιτείε. Ε, λοιπόν, θα αποχωρήσουν οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών και το τελευταίο διάστημα, δύο χρόνια, έχουμε κάνει πολλές προσπάθειες για την εκπαίδευση του στρατού και περίπου στο 99% των διαφόρων δράσεων διεξάγονται από τις Ιρακινές ένοπλες δυνάμεις. Βεβαίω αυτό που μας λείπει ε, είναι η αεροπορία. Ε, μας καλύπτουν οι Αμερικανοί προς το παρόν για την πολεμική αεροπορία, αλλά σιγά σιγά θα αποκτήσουμε και αεροπορία. Το πρόβλημα των προσφύγων είναι πάρα πολύ οξύ και σοβαρό πρόβλημα. Και μάλιστα ανθρωπιστική φύσεως. το Ιράκ δεν έχει παράδοση ως χώρα εξαγωγής προσφύγων ή παραγωγής προσφύγων. Το αντίθετο. Ε, δεχτήκαμε εκατομμύρια Αιγυπτίων στη δεκαετία του 80. Είναι μια χώρα πλούσια. Αλλά μετά από όλους αυτούς τους πολέμους που ζήσαμε και την απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας θυμάστε ότι ήμασταν υπό μποϊκότ και ξεκίνησε η διαρροή εγκεφάλων τότε. Εδώ να δείτε στο Βέλγιο είναι πολύ Ιρακινοί και στην Ευρώπη που ήρθαν ως οικονομικοί μετανάστες. Ορισμένοι και πολιτικοί, αλλά περισσότεροι οικονομικοί μετανάστες. Και μετά το 2003, τις επιθεσεις Αλ τα κτλ. Ε, το Ιράκ ήταν στα πρόθυρα στο χείλος του εμφυλίου πολέμου. Και άρχισε η βία μεταξύ των διαφόρων ομάδων και θρησκειών και πολλοί ε, διέφυγαν προς γειτονικές χώρες, Συρία, Ιράν, την Ιορδανία, την Αίγυπτο και το Λίβανο. Τώρα δίστανται απόψεις για τους αριθμούς. Οι γειτονικέ κυβερνήσει μα λέγουν ότι είναι πάνω από ένα εκατομμύριο, μία μισό εκατομμύριο άλλοι. Ε, η ύπατη αρμοστία του για του πρόσφυγε λένε ότι είναι 220.000 Ιρακινοί μόνο που έχουν καταγραφεί ω πρόσφυγε. Ιρακινοί. Σιγά σιγά Όσο βελτιώνεται η κατάσταση, οι Ιρακινοί βγαίνουν από τη χώρα, αλλά δεν είναι πρόσφυγες, είναι τουρίστες και στην Ευρώπη έρχονται ταξίδι. Επιστρέφουν στη χώρα δηλαδή, ταξιδεύουν οι άνθρωποι. Ε, και θέλω να ευχαριστήσω τις χώρες που τις υποδέχτηκαν, τους Ιρακινού αυτούς και τους προσέφεραν πολύ μεγάλη υποστήριξη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν πάρα πολύ γενναιόδορη σε αυτή την προσπάθεια. σχηματισμό κυβέρνηση. Α, προς το παρόν νόμιζα ότι ρωτούσατε για το Βέλγιο. Ε, είναι περίπλοκο. Είχαμε μια δικτατορία στο παρελθόν και μετά από τη δικτατορία, μάλλον σε περιόδους δικτατορίας, είναι εύκολο σχηματίσει κυβέρνηση. Σε ένα λεπτό αποφασίζει ο Σαντάμ και διορίζει. Τώρα δεν είναι εύκολο ο σχηματισμός κυβέρνησης. Για παράδειγμα, στην, αρχή, στην προηγούμενη κυβέρνηση οι Σουνίτες μποϊκόταραν τις εκλογές. Και τώρα οι Σουνίτες που είναι μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού συμμετείχαν σε εκλογέ, το ποσοστό 62% κάτι τέτοιο. Για πρώτη φορά οι Ιρακινοί ενώνονται, αρχίζουν να διαπραγματεύονται. Είναι πολύ μεγάλη η καχυποψία που επικρατεί ακόμα. Είναι γεγονός και θα πρέπει να μάθουμε να εμπιστευόμαστε ένα τον άλλο, να ακούμε ένα τον άλλο, να δεχόμαστε τον άλλο, να κάνουμε συμβιβασμούς, να κάνουμε διάλογο. Αυτά είναι μπροστά μας ακόμα και γίνονται σιγά σιγά ε, συγκροτημένες προσπάθειες που θα καρποφορήσουν στο τέλος. Λίγη υπομονή χρειάζεται. Κυρία Γκόμες. Okay. Oh, yes. Yeah, this is the problem. Intervention of neighboring country αυτό είναι πρόβλημα, ναι. Επέμβαση γειτονικών κρατών. Κοίτα, το γείτονά σου ούτε τον διαλέγεις ούτε τον αλλάζεις. Και στο Ιράκ το ίδιο ισχύει. Και είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση αυτή. Και πριν το 2003 είχαμε πολύ κακές σχέσεις με τους γείτονες. Εισβάλαμε στο Κουβέιτ το 80, είχαμε πολέμους με το Ιράν και με τη Συρία είχαμε δυσκολίες. Το ίδιο κόμμα, Μπαθ, αλλά με διαφορετικά καθεστώτα και ήταν αδελφά κόμματα μεν, αλλά σε εχθρική σχέση μεταξύ τους. Για να είμαι ειλικρινής, ήταν πολύ μεγάλα τα κενά. Όταν έπεσε ο Σαντάμ δεν έπεσε μόνο το καθεστώς, κατέρευσε όλο το κράτος. Για μήνες δεν υπήρχε ούτε ένας αστυνομικός, πουθενά. Και δεν ξέρουμε, ούτε τροχονόμος. Περίεργο πράγμα πώς ε, υπήρχε και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων. Και όταν υπάρχει ένα κενό, το κενό κάποιο έρχεται να το καλύψει. Και ήρθαν κάποιοι γείτονέ μα να το καλύψουν και διήρκησε αρκετό διάστημα και είναι κρίμα που οι Άραβες αδερφοί μας που θα έπρεπε να είναι εκεί πριν από όλους που έχουν κοινά πολλά μαζί μας και κοινά συμφέροντα δεν ήρθαν και μερικές ε, από τις βασικές αραβικές χώρες ακόμα απουσιάζουν και μέμφονται άλλες χώρες γιατί επεμβαίνουν. Ας επέμβουν και αυτές. Γιατί δεν το έκαναν. Και στις τελευταίες εκλογές ήταν περιφερειακές εκλογές θα έλεγε κανείς, όχι μόνο του Ιράκ, για να είμαι ειλικρινής και off the record. Επεμβαίνουν όλοι οι γειτονέ μας, μεγάλοι, μικροί, όλοι, με διάφορους τρόπους και για διάφορους λόγους. Η δημοκρατία ε, στην περιοχή δεν είναι ευπρόσδοξη. Είναι πονοκέφαλος για πολλές χώρες. Και όλοι θέλουν να φτιάξουν το Ιράκ σύμφωνα με τις δικές τους επιθυμίες και συμφέροντα είναι η δεύτερη μεγαλύτερη χώρα σε αποθεματικά πετρελαίου. Δύο εκατομμύρια βαρέλια τη μέρα. Υπογράψαμε σημαντικές ε, συμφωνίες και συμβάσεις με μεγάλες εταιρείες και τώρα θα είμαστε σε θέση να εξάγουμε 6 με 10 εκατομμύρια βαρέλια σε 10 χρόνια. Σε 6 χρόνια, συγγνώμη. Ε, δεν θα χαρούν και πάρα πολλέ γειτονικέ χώρε από αυτή την εξέλιξη, αλλά προσπαθούμε αν τι άλλο. Δεν θέλουμε να επεμβαίνουμε εμεί στου γειτονέ μα, προσπαθούμε να έχουμε διάλογο και να του πείσουμε ότι το καλύτερο και για μα και για την περιοχή και για τον κόσμο όλο. Ε, είναι αυτό. Γιατί η περιφέρεια είναι από τις πιο πλούσιες σε πηγές ενέργειας και θα πρέπει να επικρατεί ασφάλεια και ειρήνη. Είναι εκ των όνων κάλεφ για τον υπόλοιπο κόσμο και για την Ευρώπη ε, την ίδια και θα πρέπει να έχουμε οικονομική συνεργασία με ολοκληρωμένες οικονομίες. Πιέζουμε πάρα πολύ γι' αυτό. Ε, Κυρία Γκόμες, ρωτήστε για τους εσωτερικά εκτοπισμένους και αυτό είναι άλλη όψη του νομίσματος των προσφύγων. Όταν άρχισε ε, η αντιπαλότητα μεταξύ των διαφόρων θρησκευτικών ομάδων, Έφυγε ο κόσμος από τα σπίτια του, εγκατέλειψε τις αιστείες του και οι Σιήτες και οι Σουνίτες για να συγκεντρωθούν μεταξύ τους, να πάνε εκεί που ήταν οι υπόλοιποι. Αυτό συμβαίνει. Ξέρετε, και είναι η τελευταία φάση της εθνικής συμφιλίωσης, η επιστροφή των εσωτερικά εκτοπισμένων. Πολλοί επέστρεψαν. Εγώ ήμουν στις Βρυξέλλες, αλλά αν ήμουν στο Ιράκ δεν θα μπορούσα να πάω να δω το σπίτι μου. Αλλά μου λένε τώρα οι γείτονέ μου ότι έχουν αλλάξει τα πράγματα. Υπάρχουν όμως ακόμα περιοχές που έγινε εθνοκάθαρση και πολύ. Ε, αυτή σταδιακά θα αποκατασταθεί η ομαλότητα, αλλά προς το τέλος της συμφιλίωσης. NGOs, uh, ε, ε, μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Κυρία Γκόμες, τι είναι αυτά, ε, ανθρώπινα δικαιώματα. Προσπαθώ να περιοριστώ χρονικά. Αυτό δεν ήταν στο λεξιλόγιό μας. Οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις, τι είναι αυτό, ανθρώπινα δικαιώματα. Ούτε δορυφόρο είχαμε, ούτε κινητά τηλέφωνα, ήμασταν αποκομμένοι από τον υπόλοιπο κόσμο. Σιγά σιγά αρχίζουν αυτά να στείνονται. Βεβαίω υπάρχουν παραβιάσει ανθρωπίνων δικαιωμάτων και είναι δύσκολο. Αλλά έχουμε Υπουργείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Και προσεχώ θα έχουμε και ανεξάρτητη επιτροπή για ανθρώπινα δικαιώματα από την κυβέρνηση. Η τελευταία έκθεση που δημοσιεύτηκε πριν από τρεις μέρες από τον ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα βασίζεται μόνο στην πληροφόρηση ε, για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Καλό είναι αυτό, αλλά ακόμα απομένουν πολλά να γίνουν. Είναι νέα αυτά τα στοιχεία για μας και μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Όταν πρωτοεφανίστηκαν ήταν πολύ εύκολη διαφθορά. Και πάλι στο πλαίσιο αυτό που λειτουργούν. Πάντως τώρα νομίζω ότι είναι πολλές ε, οι ΜΚΟ που εργάζονται στο Ιράκ και πιέζουν και ο ρόλος τους αυξάνεται. The framework, the MOU energy and the ACAS. Yes, it was... Το πλαίσιο για την ενέργεια και τα ευρωπηγές της ΟΚΑΠ. Ναι, ήταν σημαντικό αυτό. Υπήρξε ένα είδος συμφωνίας και νομίζω και οι δύο πλευρέ, και το Ιράκ και η Ευρωπαϊκή Ένωση με τη Γενική Διεθνή Ενέργεια, εργάστηκαν ενεργά για το θέμα αυτό και ήταν ιδιαίτερα ενθουσιώδης. Εμεί σα χρειαζόμαστε, χρειαζόμαστε την Ευρωπαϊκή Ένωση και όλοι συνειδητοποιούμε τι δυσκολίε έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να διαφοροποιήσει τι πηγέ από τι οποίε προμηθεύεται ενέργεια. Εμείς είμαστε παραγωγοί Οπότε είναι αμοιβαίως συμφέρουσα και για τις δύο πλευρές η συμφωνία. Σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο, νομίζω έχουμε υπογράψει ήδη κάτι και για το φυσικό αέριο. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να αρχίσουν δημοτεύσεις τεχνικού περιεχομένου μεταξύ ΡΑΚ και Επιτροπής Ενέργειας. Για να πάρει σέρκα και ο αυτό το μνημόνιο συνεννόησης και η όλη συμφωνία για το πετρέλαιο και το φυσικό Τώρα για την κεντρική περιοχή. Είμαστε μια ομόσπονδη χώρα. Έχουμε ένα κεντρικό σύνταγμα, ομοσπονδιακό, και έχουμε και κεντρική περιοχή, έχουμε την περιοχή πίσω στο Κουρδιστάν, στα βόρεια της χώρας. Αυτή είναι και η μας, αυτός είναι ο δικός μας πολιτισμός, η δική μας κουλτούρα. Κάποιοι πιστεύουν ότι υπάρχει κεντρικός χαρακτήρας. Κάποιοι ερμηνεύουν οποιαδήποτε τάση ομοσπονδιακή ως ε, αποσχιστική. Πολλές φορές βλέπουμε και το Βέλγιο ως παράδειγμα κράτους οργανωμένου έτσι. Ναι, υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν δυσκολίες και παρανοήσεις μεταξύ κεντρικής κυβέρνησης και περιφερειακών κυβερνήσεων. Όμως, νομίζω ότι προς όφελος και των δύο πλευρών μπορούμε να βρούμε συμφωνία. Υπήρχαν πολλά, πολλά διέξοδα, το ζήτημα του Κυρκούκ είναι σημαντικό. Το Σύνταγμα όμω ε, προβλέπει κάποια πράγματα και υπάρχει οδικός χάρτης, χάρτης πορείας. Είναι σημαντικό λοιπόν οι περιφέρειες στο Ιράκ, οι επαρχίες. Είναι ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του Ιράκ και νομίζω ότι τα πράγματα οδηγούνται προς μια αρμονική επίλυση. Το Κουρδιστάν είναι σημαντικό, είναι μέρος του Ιράκ. Είναι λοιπόν προς όφελος και των Ιρακινών να επιληθεί οποιοδήποτε ζήτημα. Κυρία Πρόεδρε, Λόκπιλερ πρόεδρε τη αντιπροσωπεία για τη σχέση με το Ιράν. Σα ευχαριστώ για την ερώτησή σα. Τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Ιράν. Όπω εξήγησα νωρίτερα, αυτό για μα είναι κάτι τελείω καινούριο. Έχουμε όμω τώρα ένα Υπουργείο, έχουμε μια εξαιρετική Υπουργό. Είναι χριστιανή και είναι πολύ ειλικρινή. Και λέει ότι πάντοτε θα έχουμε κάποιε δυσκολίε και στα Υπουργεία και στην κυβέρνηση. Όμω έχει πολύ στήριξη και από το Κοινοβούλιο και από τι μη κυβερνητικέ οργανώσει και γενικώ από το κοινό λόγω χάρη τα βασανιστήρια. Ναι, κάτι τέτοιο μπορούμε να πούμε ότι διαπιστώθηκε και όχι μόνο στις δυτικές μας φυλακές και κατά τη διάρκεια της αμερικανικής κατοχής. Αλλά κατά τη διάρκεια εγκαθίδρυσης μιας δημοκρατίας υπάρχουν τέτοιου είδους συμπεριφορές. Ξέρω ότι αυτό δεν θα έπρεπε να συμβαίνει. Ε, αναφέρατε φυλακισμένους. Όμως τώρα κανείς δεν μπορεί να κρατείται εάν δεν υπάρχει δικαστική απόφαση. Και αυτή είναι μια τάση που ενισχύεται καθημερινά, με το μήνα. Δεν είναι τα πράγματα σήμερα όπως πέρσι. Ούτε όπως ήταν πριν δύο και τέσσερα χρόνια. Κινούνται τα πράγματα. Όμως, το ότι κινούνται αργά δεν θα πρέπει να μας αποθαρρύνει ούτε εμάς οποιονδήποτε θέλει να φροντίσει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Επίσης, ναι, έχει κατασταλεί η ελευθερία, ιδίω του τύπου. Τώρα όμως την αποκαταστήσαμε Α, και είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Έχουμε πλέον εφημερίδες, μία για την ε, κυβέρνηση και μία για την αντιπολίτευση, το ίδιο και με τους ραδιοφωνικούς σταθμούς. Υπάρχουν πολλές εφημερίδες φωνητικές και κανένας δεν τους ελέγχει. Βεβαίως αν υπάρχει κάποια κατηγορία μπορεί κανείς να προσφύγει στη δικαιοσύνη. Υπάρχει αυτή η διαδικασία. Συνέβη λοιπόν και αυτό. Υπήρξαν φυλακίσεις, υπήρξαν δολοφονίες, όμως σε κάθε περίπτωση τα πράγματα αποκαθίστονται, έστω και αργά. Μετά από 35 χρόνια βίαιου δικτατορικού καθεστώτος, δεν είναι εύκολο Συμφωνώ μαζί σα. Δεν πρέπει να υπάρχει καμία κακομεταχείριση βεβαίω. Πρέπει να πάψουν τελείω τέτοια φαινόμενα. Επίσης, είδαμε η Μουτζαχεντίνα ήταν οι Μουτζαχεντίν του λαού να είναι υποστηρικτέ του Σαντάμ και να είναι οργανωμένοι και σε συγκεκριμένη περιοχή. Τους βλέπαμε και στην τηλεόραση. Και υπήρχαν υποστηρικτέ του Σαντάμ που φράζονταν ελεύθερα στην τηλεόραση. Ο, η κυρία Και ακούσαμε για δολάρια που τυλίγονταν σε εφημερίδες για να διακινηθούν. Ακούσαμε τι έγινε με τους γονείς όσων έχασαν τη ζωή τους. Ε, αλλά δεν έχουν ε, πάθει τίποτα πλέον Κανείς δεν τους πειράζει. Ε, μιλάμε για την επικράτεια του Ιράκ. Σε μερικά σημεία δεν γνωρίζουμε καθόλου τι συμβαίνει. Κάποιοι έχουν να αντιμετωπίσουν ενεργούς υποστηρικτές, παθιασμένους, φαρατισμένους υποστηρικτές και δεν μπορούν ε, επίσης να αναγκαστούν να φύγουν από το Ιράκ. Δεν μπορούμε να τους στείλουμε με το ζόρι πίσω στο Ιράν. Υπάρχουν ε, γονείς, μητέρες, παιδιά, είναι 3.000 κάποιοι έχουν αμερικανικό, ευρωπαϊκό, καναδέζικο διαβατήριο. Γιατί να μην πάνε πίσω στη χώρα του, θα πει κανεί. <clears throat> γιατί δεν μπορούμε να τους υποχρεώσουμε να πάνε στο Ιράν, αν και δεν τους θέλουμε. Μπορεί βεβαίως με δικαστική κλήταξη να πάνε σε ένα δικαστήριο. Εκεί μπορούν να προσεχθούν, να προσεχθούν στη δικαιοσύνη. Όμως κάποιες φορές έχουν και στοιχεία που μπορούν να επιτελεστούν και νομίζω ότι μια τέτοια υπόθεση εκδικάστηκε χθε ή προχθέ. Πρόεδρο, ευχαριστούμε. Ο χρόνο περνάει γρήγορα. Έχουμε ακόμη τέσσερι αγορητέ. Να παραμείνουμε στο 1,5 λεπτό για τον καθένα. Κύριο Μάγερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας προτείνω για επόμενες συζητήσεις, για να μην έχουμε κατηγορίες βουλευτών πρώτης και δεύτερης κατηγορίας, να μοιράσουμε το χρόνο σε όλους και όχι να μοιρούν ε, πολύ ε, και άλλοι λιγότερο. Κύριε Πρέσβη, και εγώ εξεπλάγην από τις δηλώσεις του Πρόεδρου της Αντιπροσωπείας που είπε ότι φοβάται ότι μπορεί το Ιράν να επιβάλλει πρωθυπουργό αχυράνθρωπό του. Πραγματικά εξεπλάγει. Γιατί σύμφωνα με τη στρατιωτική ε, θεωρία, αυτός που έχει επιρροή είναι εκείνος που κατέχει έδαφος. Και έδαφος κατέχουν οι Αμερικανοί τώρα με 100.000 και πλέον στρατιώτες. Τι είναι αυτά, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στις δηλώσεις. Η Αλληρακία και η Εθνική Ιρακινή Συμμαχία ε, έχουν καταγγείλει νοθεία στις εκλογές για ακύρωση και απόσυρση 52 υποψηφίων που συνδέονται με το ΠΑΘ από ό,τι ακούγεται και μπορείτε να μας πείτε αν σε αυτή την κατάσταση που είναι τόσο δύσκολη να σχηματιστεί κυβέρνηση ε, αν δεν επηρεάζει και το Σύνταγμα που είναι θρησκευτικό και κατανέμει ότι θα πρέπει να είναι Σίτη ο Πρωθυπουργό Σουνίτη, ή κούρδο ο Πρόεδρο. Δεν ξέρω σε αυτή την κατανομή που είναι από το ίδιο σα το Σύνταγμα υπάρχει κάποια δυσκολία. Και τελειώνω για να τηρήσω και το λεπτό μου. Η δική μου πολιτική ομάδα ανέκαθεν ήταν κατά τη εισβολή. Είναι παράνομο αυτό ο πόλεμο που έφερε μεγαλύτερη ε, αβεβαιότητα ούτε τάξη έβαλε, ούτε αρακάιντα υπήρχε, ούτε ε, μέσα μαζικής καταστροφής, πετρέλαιο υπήρχε. Και σας ρωτάω για το πετρέλαιο, γιατί ήταν το πραγματικό συμφέρον στον πόλεμο του Ιράκ. Από ό,τι φαίνεται, καταφέρατε από την Ιαπωνία ένα τρεις δολάρια, συγγνώμη, ένα δολάρια για να... Ε, ε, εξυγχρονίσετε τη βασόρα και σας λείπουν άλλα 9 με 10 δις για να ε, εξυγχρονίσετε και την εξόριξη για να επανέλθετε σε επίπεδα ε, προπολεμικά. Ευχαριστώ. Κύριος Κατσίν. Ε, Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Μεσοποταμία το Ιράκ δηλαδή είναι σύμβολο, είναι κοιτίδα του πολιτισμού, είναι σύμβολο για την πολυγλωσία και για την πολυ... πολιτισμικότητα. Τώρα το Ιράκ είναι νέο κράτος και θα πρέπει να δημιουργηθούν νέοι θεσμοί και χρειάζονται χρόνο. Και καλό είναι να χρειαστεί ο χρόνος. Χωλαίνει όμως η σύγκριση με το Βέλγιο, γιατί το Βέλγιο έχει βασιλιά που εκπροσωπεί το κράτος. Ε, όμως στο Ιράκ δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Χρειάζεστε πρόεδρο, ε, βουλή και κυβέρνηση. Και ένα θετικό μήνυμα να βγαίνει από τη χώρα. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλουμε να έχουμε ισορροπημένες σχέσεις με ε, όλο σας το Κοινοβούλιο και όλη τη χώρα. Στο μέλλον θα προσπαθήσουμε να αποφύγουμε άχρηστα επεισόδια σαν αυτά που ζήσαμε πρόσφατα. Θέλουμε καλή σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το σύνολο του Ιράκ. Προσωπικά έχω πάει στο Ιράκ, στο Κουρδιστάν βέβαια μόνο. Θα πρέπει οπωσδήποτε να σχηματιστεί η κυβέρνηση έτσι ώστε το σύνολο της χώρας να ανοίξει για επισκέψεις ε, ξένων τουριστών και η Βαγδάτη να ανακάμψει η οικονομία. Γι' αυτό σας ρωτώ κύριε ε, Πρέσβη πώς σκοπεύει η χώρα να ανανεώσει τις υποδομές και ενέργειας και μεταφορών και τι θέλετε να κάνετε για την ανάπτυξη της οικονομίας. Μετά από τόσα χρόνια πόλεμο δεν έχει έρθει η ώρα να ανανεωθεί η χώρα. Με συναρπάζει και το δυναμικό και οι δυνατότητες της γεωργίας στη Μεσοποταμία. Ξέρετε τι δυνατότητες έχετε. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ράτκινς. Πάντοτε είμαι σύντομο, κύριε Πρόεδρε. Έχω δύο σύντομα ερωτήματα. Πρώτον, για τι υποδομέ, ιδίω μετά από μια προηγούμενη ερώτηση. Τι συμβαίνει σε σχέση με το επίπεδο κεντρικής κυβέρνηση κυβέρνησης και περιφερειακών κυβερνήσεων, ιδίως όσον αφορά τις υποδομές για την ηλεκτρική ενέργεια. Δεύτερον, τι συμβαίνει για την προστασία των αρχαιοτήτων. Υπάρχει μεγάλος αριθμός αρχαιοτήτων στη χώρα σας και πολύ ανησυχούμε για την τύχη τους. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρος. Ο κύριος Τάνοκ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε έχω κάποιες ερωτήσεις. Καταρχήν, όλοι αναγνωρίζουμε ότι η ομοσπονδιακή δομή του Ιράκ είναι πολύ ευάλωτη. Αυτό, κατά τη γνώμη του πρέσβη, ε, είναι πολύ πολιτικό βέβαια το θέμα για να το απαντήσει ένας πρέσβης. Ε, θεωρείτε ότι αυτό σημαίνει ε, ότι μπορεί να υπάρχει ένας μόνιμος συνασπισμός που θα συμπεριλαμβάνει και τους Σουνίτες ή μπορεί να ισχύσει μια ομοσπονδιακή μορφή που θα υπάρχει πλειοψηφία Σιητών και μειοψηφία Σουνιτών με ενδιαφέρει ιδιαίτερα το θέμα των διμερών σχέσεων μεταξύ του Ιράκ και των Αράβων γειτόνων του, ιδίως με τη Σαουδική Αραβία που ανησυχεί για την επιρροή του Ιράν στην Βαγδάτη και επίσης με τη Συρία για τους αντίθετους λόγους ότι επειδή υπάρχει στενή σχέση Δαμασκού και Τεχεράνης είναι το μόνο επιζών καθεστώς ε, Μπαφ ε, θέλει να έχει καλές σχέσεις ε, στο μέλλον με τη νέα κυβέρνηση στη Βαγδάτη. άλλο ένα ερώτημα που με ενδιαφέρει πάρα πολύ στο Ηνωμένο Βασίλειο εγώ είμαι ε, μεταξύ των υποστηρικτών της οργάνωσης ε, για την ε, διάσωση των ασυρίων και των Ασυριακών μνημείων και αναφέρθηκαν τα μνημεία, αλλά τι θα γίνει με τους ασυρίους που διέφυγαν από τη χώρα. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω σας δώσω 5 λεπτά, κύριε Πρέσβη, για να μπορέσετε να απαντήσετε. Σας δίνω λιγότερο χρόνο, ίσως είναι προς όφελό σας. για την ερώτηση του κ. Μάγερ για την προσπάθεια ε, επιβολή κυβέρνηση από το Ιράν στο Ιράκ. Δεν νομίζω ότι είναι δυνατόν αυτό. Είχαμε ε, ελεύθερε εκλογέ, υπήρχαν κάποιε δυσκολίε, αλλά όχι σε τέτοιο βαθμό. Και μεταξύ μας ε, αυτοί που κατηγορούνται ότι πρόσκυνται στο Ιράν δεν είναι και κάποιοι που κέρδισαν ε, πάρα πολλές, ψήφου. ψήφους θα είναι μια κυβέρνηση πολυσυλλεκτική και αντιπροσωπευτική όλων των συνιστοσών της κοινωνίας του Ιράκ και Σιητών και Σουνιτών και Κούρδων και Τουρκμένων. Έτσι πρέπει να είναι και έτσι θα είναι, είναι η μόνη λύση. Και όλοι οι πολιτικοί το αντιλαμβάνονται και είναι ο μόνος τρόπος κατά τον οποίο μπορεί να δημιουργηθεί μια νέα κυβέρνηση και γι' αυτό και παίρνει πολύ χρόνο ο σχηματισμός της νέας κυβέρνησης. Δεν θα είναι ούτε ΣΥΙΤΕΣ, ούτε Σουνίτες, ούτε στο Σύνταγμα υπάρχει κάτι από αυτού. Οι σύντες είναι η πλειοψηφία. Κατά πάσα πιθανότητα θα έχουν λοιπόν επαρκή πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο και θα τα συμφωνήσουν μεταξύ τους. Δεν έχουν ακόμη συμφωνήσει μεταξύ τους. Αλλά δεν θα πρέπει να μας εκπλήσει αν ο επόμενος Πρωθυπουργό είναι Σίτη. Αλλά ο μόνος λόγος είναι ότι αυτό είναι αποτέλεσμα δημοκρατικής διαδικασίας. Όσον αφορά το πετρέλαιο. Πριν από λίγου μήνε, το Ιράκ υπέγραψε μεγάλε συμφωνίε ε, με σημαντικέ πετρελαϊκέ εταιρείε και οι περισσότερε είναι ευρωπαϊκέ, πρέπει να πούμε. Οι Αμερικανοί πήραν μια μικρή σύμβαση. Ένα μικρό μερίδιο σε μια σύμβαση. Δεν θα έπρεπε λοιπόν να ανησυχείτε. Όσον αφορά τις σχέσεις ε, μεταξύ της Ιρακινής Βουλής των Αντιπροσώπων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ε, συμφωνώ πλήρως. Ε, τώρα έχουμε ένα νέο κοινοβούλιο, δεν έχει ακόμη συγκληθεί για να εκλέξει τον πρόεδρό του, αλλά μόλις εκλέξει και πρόεδρο και συγκληθεί, νομίζω ότι θα πρέπει να ξεκινήσουμε αμέσω τις σχέσεις. Και βλέπω και τον κύριο Πέτερινγκ εδώ. Όταν ήταν πρόεδρος, ο κύριος Πέτερινγκ μας υποστήριξε πάρα πολύ και σας ευχαριστώ κύριε Πέτερινγκ, χαίρομαι που σας βλέπω. Τώρα, επενδύσεις και ανάπτυξη και σχετικά προγράμματα. Όντως, χρειαζόμαστε επενδύσεις και δεν έχουμε πολλές δυνατότητες και το Κοινοβούλιο ψήφισε ένα ιδιαίτερα ενθαρρυντικό νόμο για τις επενδύσεις και τώρα περιμένουμε τις επενδύσεις. Έρχονται επενδύσεις από τη Γαλλία, από την Κίνα. Οι Κινέζοι είναι οι πρώτοι που έρχονται πάντοτε. Από την Τουρκία, κάποιες βελγικές εταιρείες, έρχονται κάποιες γερμανικές εταιρείες. Ιδίως στον τομέα του πετρελαίου, δεν χρειαζόμαστε 10 και 15 που είπε κάποιο ευρωβουλευτή. Χρειαζόμαστε δισεκατομμύρια, εκατοντάδε δισεκατομμυρίων δολαρίων. Και σιγά σιγά έρχονται αυτέ οι επενδύσει, γιατί το πετρέλαιο όλοι το χρειάζονται. Σχέσεις με τη Σαουδική Αραβία και τη Συρία. Εδώ θα πρέπει να είμαι διπλωματικός, δεν μπορούμε να είμαι απόλυτα ειλικρινής. Ε, όπως είπαμε, δεν έχουμε τις βέλτιστες σχέσεις με κάποιους γειτονές μας. Κάποιοι γειτονές μας κατηγορούνται ότι επιτρέπουν σε τρομοκράτες ε, να περάσουν τα σύνορα και να μπουν στη χώρα μας. Δεν χαροποίησε αυτό τους γειτονές μας, αλλά είναι γεγονός. Υπάρχει παρέμβαση στην περιοχή, κυρίως από τους γειτονέ μας. Και κάποιοι γειτονέ μας δεν είναι ικανοποιημένοι, είτε διότι ε, επικρατεί σιγά σιγά δημοκρατία στην ε, γενικότερη περιφέρεια, είτε για το Ιράκ έχει συμφωνίες με πετρελαϊκές εταιρείε και είναι το Ιράκ μεγάλη ε, χώρα παραγωγός πετρελαίου και αυτό δεν του χαροποιεί. Και φτάνω τώρα και στο θέμα των μνημείων της ανθρωπότητας που χάθηκαν. Και ήταν κρίμα γιατί τα έχασε ολόκληρη η ανθρωπότητα αυτά τα αρχαιολογικά μνημεία. Συνόδευα στο Ιράκ το Βέλγο Υπουργό που επισκέπτεται το Ιράκ και μου ζήτησε να επισκεφθούμε ένα μουσείο. Πήγα μαζί του και ένιωσα πολύ καλύτερα διότι υπήρχαν ε, σε δύο μεγάλες αίθουσες ευρήματα που είχαν έρθει και από την Αμερική και από γειτονικέ χώρες και αυτό ε, μόνο κατά το ίμιση θα μπορούσε να καλύψει αυτό το οποίο είχαμε χάσει. Πάντως, στο Ιράκ, όπου και να σκάψει κανείς, ε, θα βρει ε, κάτι. Υπάρχουν πολλά αρχαιολογικά μνημεία. Έχουμε τουλάχιστον κάτι. Δεν είχαμε τίποτα με την καταστροφή, τώρα έχουμε αρχίσει να έχουμε κάτι. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Ελπίζω η συζήτηση αυτή να απάντησε κάποιες από τις ερωτήσεις μας. Και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά, κύριε Πρέσβη. Ευχαριστώ και εγώ, κύριε Πρόεδρε. Και θα συνεχίσουμε εμείς με τον ε, Πρέσβη, κύριο Τόρβαν Μπρίλε. Yeah, okay. Don't go away. Stay put. Okay then. Well, thank you, Ambassador, for coming. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε που είστε παρόν ε, ανάμεσά μας. Θα συζητήσουμε άλλο ένα σημαντικό θέμα για μας, τις εκλογές στο Σουδάν. Αν θυμάστε πριν από λίγο καιρό είχαμε τον πρώην πρόεδρο της Αφρικής, τον κύριο Τάμπο Μπέκη και συζητήσαμε πολλά προβλήματα σε σχέση με τις επερχόμενες τότε εκλογές. Υπάρχει και το θέμα του δημοψηφίσματος για την αυτοδιάθεση στο Νότιο Σουδάν που θα διεξαχθεί τον Ιανουάριο Και θα έρθουν και δύο συνάδελφοι σε λίγο που είναι ή θα έρθουν σε λίγο. Βερονίκ Τεκάιζερ, η κυρία βερονικ τεκαιζερ Συνάδελφοι που έχουν επισκεφθεί τη χώρα. Έχετε το λόγο κύριε Πρέσβη. Ευχαριστώ. Yeah, that's uh, Mr. President, thank you very much and thank you very much to Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ όλου που μου δώσατε την ευκαιρία να πω δύο λόγια για την κατάσταση στο Σουδάν. και για την επερχόμενη περίοδο στο Σουδάν που θα είναι αποφασιστική στιγμή στην ιστορία του Σουδάν. Νομίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε τον επικεφαλής ε, της Ευρωπαϊκής ε, Αποστολής Παρατηρητών κατά τις εκλογές του Σουδάν, αλλά δεν θα σας πω εγώ τίποτα για τις, δεν θα σας δώσω λεπτομέρειες για τις εκλογές. Το μόνο που θα σας πω είναι ότι διεξήχθησαν οι εκλογές. Ε, και στην νέα κυβέρνηση οι ίδιες προσωπικότητες υπάρχουν. και συνεχίζει να ισχύει η ολοκληρωμένη ειρηνευτική συμφωνία η οποία συνήθι το 2005 μετά από 20 χρόνια εμφύλιου πολέμου στο Σουδάν και τώρα μπαίνει στην τελική και κρίσιμη φάση της. Όπως πολύ σωστά είπε ο Πρόεδρος, τον Ιανουάριο την επόμενη χρονιά θα διεξαχθεί δημοψήφισμα στο Νότιο Σουδάν, όπου ο λαός του Νοτιού Σουδάν θα αποφασίσει αν θέλει να μείνει στο ενιαίο Σουδάν ή αν θέλουν να αποσχιστούν ως ε, αυτόνομη χώρα. Μια πολύ σημαντική στιγμή λοιπόν στην ιστορία της χώρας αυτής, ε, μια αποφασιστική περίοδος ε, για ολόκληρη την περιφέρεια, γιατί το Σουδάν είναι η μεγαλύτερη γεωγραφικά χώρα στην Αφρική με σύνορα στα οποία επικρατούν ασταθείς ε, συνθήκες στις περισσότερες περιπτώσεις και για την υπόλοιπη Αφρική λοιπόν το μέλλον του Σουδάν έχει πολύ μεγάλη σημασία. Η οριστικοποίηση της ολοκληρωμένης συμφωνίας ειρήνης συμπεριλαμβάνει και το δημοψήφισμα που θα γίνει τον Ιανουάριο του 2011. Περιλαμβάνεται λοιπόν στην ειρηνευτική συμφωνία την οποία προσυπέγραψαν και οι δύο πλευρές και την οποία ε, εγγυάται η διεθνής κοινότητα. Υπάρχουν και άλλα στοιχεία στην ολοκληρωμένη ειρηνευτική συμφωνία που πρέπει ακόμη να υλοποιηθούν. Ένα κέριο σημείο είναι η οριοθέτηση των συνόρων μεταξύ Βορείου και Νοτιού Σουδάν. Προφανώς αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο, λαμβάνοντας υπόψη ότι το Νότιο Σουδάν θα ψηφίσει ως Νότιο Σουδάν και υπάρχει και το θέμα των τριών μεταβατικών ε, περιοχών ε, της περιοχής που ονομάζεται ABA μια περιοχή όπου ε, το Διεθνές Διατητικό Δικαστήριο έλαβε μια απόφαση πέρυσι σχετικά με την οριοθέτηση των συνόρων αλλά πολλά στοιχεία στην απόφαση του Διαιτητικού ε, Δικαστηρίου παραμένουν ακόμη προς απόφαση. Κάτι άλλο που είναι σημαντικό είναι το να ε, διεξαχθεί το δημοψήφισμα με τρόπο ώστε να είναι αξιόπιστο το αποτέλεσμά του. Απαιτεί λεπτομερή προετοιμασία και επίσης ε, απαιτείται τα συμβαλόμενα μέρη, τα εμπλεκόμενα μέρη ε, να αντιλαμβάνονται την αναγκαιότητα που υπάρχει να συζητήσουν τα διάφορα θέματα και ε, σίγουρα θα υπάρξουν πολλά συμπεράσματα που μπορούμε να αντλήσουμε από τις αποστολές παρατήρησης των εκλογών, μεταξύ των οποίων και η δικιά μας, συμπεράσματα που θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε για την προετοιμασία του δημοψηφίσματος. Ακόμη θα πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα τα θέματα που οι Σουδανοί ονομάζουν θέματα για μετά το δημοψήφισμα, δηλαδή θέματα που πρέπει να διαπραγματευτούν τα εμπλεκόμενα μέρη για να διασφαλιστεί ειρηνική συνύπαρξη ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος στο Νότιο Σουδάν. Τα θέματα τα οποία συμπεριλαμβάνονται εδώ είναι η ασφάλεια, η ηθαγένεια, τα θέματα των ε, οικονομικών και φυσικών πόρων, διεθνείς συνθήκες. Ευτυχώς πρόσφατα, κατά τη σύνδεση μιας συμφωνίας μεταξύ των δύο μερών στην Αιθιοπία, στο Μακέλε, υπεγράφει ένα μνημόνιο συνεργασίας ε, μεταξύ ε, των ε, δύο επικεφαλής των διαπραγματεύσεων και αυτό το μνημόνιο συνεργασίας σαφώς δηλώνει ότι θα πρέπει τα δύο, τα δύο εμπλεκόμενα μέρη να αναλάβουν αυτή τη διαδικασία, αλλά ίσως να χρειαστεί και κάποια διευκόλυνση, κάποια μεσολάβηση και αναφέρεται και ε, Αφρικανική Ένωση και ίσως ο, πρόεδρος, ο πρώην πρόεδρος κ. Μπέκη που αναφέρεται προηγουμένως θα είναι αρμόδιος ε, για να διευκολύνει τα εμπλεκόμενα μέρη κατά τις διαπραγματεύσεις που θα έχουν μεγάλη σημασία για τη διατήρηση ειρηνικών σχέσεων μεταξύ των δύο μερών. Η κατάσταση στο Νότο συχνά αποτέλεσε πηγή ανησυχία και πέρυσι υπήρξαν αρκετά θύματα ε, λόγω εθνοτικών διανέξεων και σειράξεων στο Νότο με προβλήματα ε, σημαντικότερα από ότι στο Νταρφούρ και υπήρξαν προβλήματα αποσταθεροποίησης ορισμένων περιοχών ελλείψεις ειδών διατροφής, ένα εκρηκτικό μείγμα σε όλη αυτή την περιοχή. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Νότος δεν είναι σε θέση να ξεπεράσει ορισμένα από αυτά τα προβλήματα, παρότι θα χρειαστεί και την υποστήριξη της διεθνούς κοινότητας και θα χρειαστεί και μια σταθερή και επικοδομητική σχέση με το Βόρειο Σουδάν. Η κατάσταση στο Νταρφούρ παραμένει πηγή ανησυχίας. Έχει επιδεινωθεί η κατάσταση ως προς την ασφάλεια της περιοχής τους τελευταίους έξι μήνες και έχουν γίνει και επιθέσεις ε, κατά της ειρηνευτικής δύναμης, ε, της δύναμης UNAMID των Ηνωμένων Εθνών. Ε, είχαμε αρκετά θύματα και οι ανθρωπιστικές επιχειρήσεις έχουν εμποδιστεί λόγω της έλλειψης πρόσβασης σε ορισμένες περιοχές όπου είχαμε ε, σειράξεις μεταξύ κυβερνητικών δυνάμεων και ένοπλων δυνάμεων και ε, σε ορισμένες περιπτώσεις επλήγησαν άμεσα οι ανθρωπιστικές δυνάμεις, οι εργαζόμενοι στις ανθρωπιστικές δυνάμεις και τρεις όμοιροι ε, παραμένουν όμοιροι, χωρίς να ε, ξέρω αυτή τη στιγμή είναι ποια είναι η δύναμη για την οποία μιλάμε, αλλά σαφώς ε, αυτό έχει επίπτωση στην δυνατότητα των ε, ειρηνευτικών δυνάμεων να επιτελέσουν το έργο τους. Στην Νιέλα, σε μια πόλη του φού σαφώς υπήρξαν τέτοια συμβάντα και εγώ ίδιος ήμουν μάρτυρας και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι οι ειρηνευτικές δυνάμεις δεν μπορούν να έχουν ελεύθερη πρόσβαση στα σημεία στα οποία θα ήθελαν να φτάσουν και οι ανθρωπιστικές επιχειρήσεις δεν μπορούν να φτάσουν σε κάποιες ε, περιοχές και ιδίως στις περιοχές όπου θα είχαν ε, την ε, μεγαλύτερη ε, σημασία και αποτελεσματικότητα. Η επίλυση δεν μπορεί να επέλθει με στρατιωτικά μέσα. Χρειάζεται μια πολιτική λύση και ένα κοινό μεσολαβητή ε, Αφρικανική Ένωση και Ηνωμένων Εθνών ε, ε, στην Τόχα κινείται προ αυτήν την κατεύθυνση και οι εκπρόσωποι τη κοινωνία των πολιτών συναντήθηκαν στην Τόχα και εγώ ήμουν παρόν για να συμμετάσχω στα, στην έναρξη ενό φόρουμ της κοινωνίας των πολιτών με στόχο να ακούγεται η φωνή των ίδιων των πολιτών στην προσπάθεια επίτευξης μιας συμφωνίας. Ξέρουμε ότι ε, κάποιοι δεν δέχτηκαν να συμμετάσχουν σε αυτές τις διαπραγματεύσεις και είναι πολύ πλοκή η κατάσταση και υπάρχει άμεση ανησυχία για θέματα ασφάλειας ε, και γιατί και ε, επικρατεί ατιμορρησία ως γενικός κανόνας και είναι απαραίτητο και η κυβέρνηση και η UNAMID να αντιμετωπίσουν αυτά τα προβλήματα. Είναι πολύ σοβαρή η κατάσταση και αυτό φαίνεται και από μια ανακοίνωση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου ότι προστίθεται άλλη μια υπόθεση ε, στις ήδη φυστάμενες καταγγελίες κατά του Προέδρου του Σουδάν. Το Νταρφούρ λοιπόν θα παραμείνει ε, ως προτεραιότητα ε, στα θέματα που μας αποσχολούν μέσα στην επερχόμενη περίοδο και θα είναι κέρια σημασία οι επόμενοι 6 έως 12 μήνες. Υπάρχουν πολλέ ανησυχίε για την κατάσταση στο Σουδάν, σε ε, ολόκληρη την ευρύτερη περιφέρεια, γιατί το Σουδάν είναι για πολλού λόγου σημαντική χώρα. Η Αφρικανική Ένωση είναι αποφασισμένη να παίξει σημαντικό ρόλο για να δημιουργηθούν ε, οι προϋποθέσεις για ειρηνική συνύπαρξη Βορρά και Νότου, ανεξάρτητα από την έκβαση του δημοψηφίσματος. Και ε, όλες οι γειτονικέ χώρες ακολουθούν την ίδια προσέγγιση. Θα πρέπει το Νότιο Σουδάν να έχει τη δυνατότητα να ασκήσει το δικαίωμα το οποίο αναφέρεται στην Ευτική Συμφωνία, δικαίωμα ψήφου λοιπόν, να αποφασίσουν αν θέλουν να παραμείνουν στο Σουδάν ή αν θέλουν να ακολουθήσουν διαφορετική πορεία Πάντω θα πρέπει να δημιουργηθούν όλες οι προϋποθέσεις ε, ούτω ώστε να υπάρχουν ε, οι συνθήκε ειρηνική συνύπαρξης που είναι απαραίτητες ανεξάρτητα με την έκβαση του δημοψηφίσματος. και όλοι οι διεθνεί φορεί θα πρέπει να φροντίσουν ε, όσο είναι δυνατόν να υπάρξει μια συνεκτική προσέγγιση στο θέμα των εξελίξεων στο Σουδάν. Θα ήθελα εδώ να αναφερθώ στη δημιουργία του Συμβουλευτικού Φόρουμ ε, από την Αφρικανική Ένωση και τα Ηνωμένα Έθνη, όπου υπάρχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι σε διεθνές επίπεδο. Και αυτό ελπίζουμε ότι θα οδηγήσει σε μια πιο συνεκτική και ολοκληρωμένη προσέγγιση στα προβλήματα του Σουδάν. Αυτά ως παρατηρήσεις προς το παρόν κύριε Πρόεδρε και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε τη συζήτηση βάσει αυτών. Σας ευχαριστώ πολύ τώρα να ζητήσω τον συνάδελφο, τον συνάδελφο, την κυρία Ντεκάιζερ, που ήταν επικεφαλής παρατηρήτρια εκ της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Σουδάν, να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητέ Τόρμπεν, με μεγάλη χαρά σε υποδεχόμεθα εδώ. Δεν ε, θα εξηγήσω όλες τις λεπτομέρειες της αποστολής στο Σουδάν. Θα δώσω απλώς ε, μια σύνθεση των αποτελεσμάτων της τελικής έκθεσης και θα μιλήσω και για το μέλλον. Πήγα στο Σουδάν πριν από 15 μέρες για να δώσω την τελική έκθεση για τις εκλογές ε, στην Επιτροπή των Εκλογών στο Βόρειο Σουδάν και πήγα επίσης και στο νότο της χώρας για να ανακοινώσω τα αποτελέσματα της έκθεσης, όχι ακολουθώντας ακριβώς την ίδια διαδικασία, για να μην βάλουμε ήδη από τώρα σε ίση μοίρα το βορρά και το νότο, σαν να είχε ήδη γίνει το δημοψήφισμα και να έχει ε, δώσει ως αποτέλεσμα την, ε, την, ε, το διαχωρισμό της χώρας σε δύο τμήματα. Είναι ιστορική σημασία σε αυτές τις στιγμές για το Σουδάν και οι εκλογές ε, ε, θεωρούνται στο Νότο, αλλά ίσως και στο Βορρά, ως υποχώρηση η οποία γίνεται ε, στην ολοκληρωμένη ειρηνευτική συμφωνία. Η ολοκληρωμένη ειρηνευτική συμφωνία που έθεσε τέλος στον πόλεμο το 2005, στον πόλεμο Βορρά Νότου, προέβλεπε διάφορα στάδια μεταξύ των οποίων οι εκλογές και το τελευταίο στάδιο είναι το δημοψήφισμα το οποίο πρέπει να διεξαχθεί τον Ιανουάριο του 2011. Όταν έγιναν οι εκλογές, στο Βορρά ε, επικράτησε μια κάπως περίεργη κατάσταση, διότι ε, όλοι οι υποψήφοι που θα μπορούσαν ε, να αντιταχθούν στον ε, πρόεδρο Αλμπασίρ με κάποια αποτελεσματικότητα ε, δεν έλαβαν ε, μέρος. Τα κύρια κόμματα της αντιπολίτευσης βοηκοτάρισαν τις εκλογές και τελικά στο Βορρά για τις προεδρικές εκλογές τουλάχιστον δεν υπήρχε νόημα γιατί υπήρχε σε γενικές γραμμές ένας μόνο υποψήφιος και δεν πρέπει να μας εκπλήσει το ότι ο Μπασίρ κέρδισε τις προεδρικές τουλάχιστον εκλογές. Βέβαια δεν υπάρχουν μόνο οι προεδρικές εκλογές, είχαμε και τις εκλογές των κυβερνητών, τις εκλογές των κοινοβουλευτικών συνελεύσεων κλπ. Παρ' όλα αυτά οι προεδρικές εκλογές ε, ε, ε, έχασαν τη σημασία του στο βαρά στο Νότο ε, είχαν υπόψη τους την ε, προοπτική του δημοψηφίσματος. Το ε, SPLM, το SPLM είναι το κυρίαρχο κόμμα, το απελευθερωτικό κίνημα των λαών του Σουδάν με τον Σαλβά Κύρ επικεφαλής και δεν θα πρέπει να σε εκπλήσει ούτε αυτό, γιατί εφόσον έχουν κατά το δημοψήφισμα, ο Σαλβά Κύρ κέρδισε τις εκλογές στο Νότο με αποτέλεσμα απόλυτα εντυπωσιακό, στα θα λέγαμε, πάνω από 92% των ψήφων. Ο Αλμπασίρ είχε την αξιοπρέπεια να περιοριστεί στο 62,8% των ψήφων. Πολύ υψηλά ποσοστά και τέθηκε το ζήτημα στην αποστολή παρατήρηση των εκλογών αν ήταν αξιόπιστα αυτά τα αποτελέσματα. Θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε διάκριση σε δύο βασικές στιγμές αυτών των εκλογών. Υπάρχει η περίοδος μέχρι τις εκλογές και η μέρα των εκλογών και μπορούμε να πούμε ότι σε γενικές γραμμές στο βορρά περισσότερο αλλά και στο νότο γενικά καλώς διαξήχθησαν οι εκλογές. Η Άννα μπορεί να ε, είναι πιο δεικτική από μένα και να σας πει ότι όχι, υπήρξε εκλογική νοθεία κλπ. Ε, ίσως να υπήρξε κάποια νοθεία που δεν την είδαμε ε, λόγω της απογραφής και ικανοποιηθήκαμε τουλάχιστον με αυτά που βλέπαμε την ημέρα των εκλογών τα οποία ήταν στο όριο μεν, αλλά πρέπει να πούμε ότι έγινε μια μεγάλη προσπάθεια. Το δεύτερο κομμάτι των εκλογών, δηλαδή το κλείσιμο των εκλογικών τμήματων. Οι εκλογέ διήρκεσαν πέντε μέρε, πρέπει να πούμε. Η καταμέτρηση, το κλείσιμο και η καταμέτρηση ήταν σε συνθήκες πανικού. Υπήρχαν 12 ψηφοδέλτια, δυσκολία στην μεταφορά των ψηφοδελτίων, πολύ μεγάλες δυσκολίες. Και αντί ε, ε, να καταχωρηθούν αυτά τα αποτελέσματα στο μηχανογραφικό σύστημα το οποίο με τη βοήθεια της διεθνούς κοινότητας είχε δημιουργηθεί για να μπορέσουμε να επαληθεύσουμε τα αποτελέσματα και να δούμε αν πραγματικά στην ΑΒ εκλογική περιφέρεια είχαμε 100% των ψήφων υπέρ ενός και μόνο υποψηφίου ή αν ε, τα ψηφοδέλτια που δόθηκαν στην είσοδο ήταν αυτά τα οποία βρίσκαμε και στην έξοδο αν υπήρχαν κάποια ψηφοδέλτια τα οποία ήταν σχισμένα αλλά έπρεπε να ληφθούν υπόψη. Αυτά που γίνονται συνήθω δηλαδή στην αναμέτρηση των εκλογών. Θα έπρεπε όλα αυτά να τα επαληθεύουμε με το μηχανογραφημένο σύστημα το οποίο είχε οργανωθεί. Η Εκλογική Επιτροπή είπε μετά από κάποιες προσπάθειες που κάνανε δεν είναι δυνατόν να μπουν στο σύστημα, το πληροφορικό σύστημα που υπάρχει, πρέπει να τα μετρήσουμε. Έκανα λοιπόν καταμέτρηση έξω από κάθε είδου παρατήρηση, πάνω σε χαρτάκια στα οποία σημείωναν. Χάθηκε λοιπόν κάθε δυνατότητα ελέγχου και επί 15 μέρες είδαμε ότι η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των προεδρικών εκλογών έγιναν με λιγότερο από 50% των ψήφων. Είπαν, α, κέρδισαν. θα μπορούσαν και να τα έχουν εφεύρει τα αποτελέσματα. Δεν ήταν δυνατόν να γίνει επαλήθευση. Δεν μπορούσαμε να ελέγξουμε τίποτα. Όλα τα συστήματα διασφάλισης διασφάλισης είχαν χαθεί και με πολύ αυστηρή παρατήρηση δεν θα μπορούσαμε να έχουμε δώσει τίποτα άλλο, δεν θα μπορούσε να υπάρχει άλλος ε, νικητής των εκλογών. Παρόλα αυτά ε, ήταν στο όριο ε, ο τρόπος ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Μπορούμε να το δούμε αυτό σαν τελευταίο βήμα προς την τελική ευθεία και προς το τελικό σημείο που είναι το δημοψήφισμα, αλλά θα πρέπει να αντλήσουμε συμπεράσματα ακριβώς για το δημοψήφισμα. Το, δημο... το δημοψήφισμα αυτό θεωρείται το μεγάλο διακύβευμα για τον Σουδανικό πληθυσμό και θα πρέπει να δούμε το τι έχει γίνει μέχρι τώρα στις ε, εκλογές αυτές. Ε, υπήρχαν ε, και περιστατικά βία στο Νότο. Είπε και ο Τόρμπεν κάτι ότι υπήρξαν κάποια ζητήματα υπήρχαν και κάποιοι από το Βορρά που ε, προσπάθησαν να δουν πώς είναι η κατάσταση στο Νότο. Δεν ήταν ιδιαίτερα δραματική η βία, αλλά η βία από τις ένοπλες δυνάμεις ή από παραστατιωτικές ε, ομάδες που μπήκαν στα εκλογικά τμήματα και που τρομοκράτησαν το προσωπικό των ε, εκλογικών τμήματων ήταν μεμονωμένα τμήματα, αλλά αν αυτό γίνει και στο δημοψήφισμα θα έχει εντελώ διαφορετική σημασία. Και αν θέλουμε να φτάσουμε στην ολοκλήρωση ε, και στην τελική ευθεία της ε, ολοκληρωμένης ε, ειρηνευτικής συμφωνίας, θα πρέπει να διδαχθούμε από αυτές τις εκλογές, και αυτό λέμε και προς τον πρόεδρο Αλ εάν ε, δεν ε, ελέγξετε την κατάσταση στο δημοψήφισμα του Ιανουαρίου, αυτό θα δημιουργήσει προβλήματα. Πρέπει λοιπόν ε, να ελέγξετε τις στρατιωτικές και παραστρατιωτικές δυνάμεις για να μπορέσετε να έχετε αξιόπιστα αποτελέσματα. Χρειάζεται πάντως οπωσδήποτε η υποστήριξη της διεθνούς κοινότητας και των Ηνωμένων Εθνών για να υπάρξει ένα ειρηνικό περιβάλλον στο οποίο θα διεξαχθεί το δημοψήφισμα. Ένα άλλο σημείο πάρα πολύ σημαντικό, στο οποίο καθυστερήσαμε πάρα πολύ, είναι το θέμα της ε, καταγραφής γιατί ε, στην καταγραφή διαπιστώσαμε πολλά σφάλματα. Δεν ήμασταν εκεί κατά την καταγραφή, αλλά διαπιστώσαμε τις συνέπειες. Τουλάχιστον 10% των εκλογέων δεν υπήρχαν του εκλογικού καταλόγους και λέω τουλάχιστον 10% γιατί αυτό έγινε μέσα στα εκλογικά τμήματα. Ε, ερχόταν κόσμο και δεν έβλεπε το όνομά του στον τοίχο, στου τυχοκολλημένου καταλόγου και ξαναέφυγαν για να πάνε να βρουν πού θα πρέπει να ψηφίσουν. Το 10% είναι μέσα στα εκλογικά τμήματα που σα αναφέρω μπορεί να υπήρξαν ε, εσφαλμένες καταχωρήσεις χωρίς να μπορούμε να το αποδείξουμε. Σε ορισμένα χωριά μπορεί να καταγράφησαν 100 άτομα που δεν ε, συμμετείχαν στην ψηφοφορία. Αν αυτό ξαναγίνει στο δημοψήφισμα, δηλαδή αν εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορέσουμε να εμποδίσουμε κάτι τέτοιο, αν κληθούμε να παρατηρήσουμε το δημοψήφισμα και δεν μπορούμε να επαληθεύουμε την ποιότητα του δημοψηφίσματος, υπάρχει μια ρήτρα για το δημοψήφισμα που έχει κέριο χαρακτήρα. Δηλαδή χρειάζεται το 60% των καταγεγραμμένων, ε, πρέπει να ψηφίσει το 60% των καταγεγραμμένων. Φανταστείτε, αν ένα κόμμα, δεν θέλω να πω ποιο κόμμα, αν ένα κόμμα θέλει να σαμποτάει το δημοψήφισμα, μπορεί να δημιουργήσει καταλόγους με ψευτοεκλογής. Μπορεί κάποιος να γράψει στον κατάλογο οικογένειες από γειτονικά χωριά που ποτέ δεν θα έρθουν να ψηφίσουν και τελικά ε, θα βγει άκυρο το δημοψήφισμα. Το θέμα λοιπόν του σωστού ελέγχου της καταγραφής των εκλογών έχει πρωταρχική σημασία. Και τα αναφέρω αυτά τα παραδείγματα διότι δηλαδή θέλω να πω ότι ε, ξέρουμε ότι ο Νότος το θέλει το δημοψήφισμα, το μεγαλύτερο μέρος ε, στο Νότο θέλει το δημοψήφισμα, αλλά όχι και όλοι. Αν αμφισβητηθεί λοιπόν η αξιοπιστία του δημοψηφίσματος και των αποτελεσμάτων του, θα είναι δραματικό. Μπορεί να υπάρξουν εντάσεις τις οποίες πρέπει να αποφύγουμε οπωσδήποτε, δημιουργώντας και ένα ειρηνικό περιβάλλον όπως είπαμε, το οποίο θα εγγυηθεί και ε, η Αφρικανική Ένωση και τα Ηνωμένα Έθνη και θα πρέπει και μια επιτροπή παρακολούθηση των εκλογών, παρατήρηση των εκλογών να διασφαλίσει τη σωστή διεξαγωγή του δημοψηφίσματος. Άλλο ένα σημαντικό σημείο που δεν ε, έχω συζητήσει ακόμη και είναι σημαντικό και θέλω να το αναφέρω είναι το εξή. Ως Επιτροπή Παρατήρησης των Εκλογών πρέπει να παρέμβουμε σε μια εκλογική διαδικασία. Έχουμε πολύ αυστηρή μεθοδολογία ε, που δεν μας επιτρέπει καμία παρέμβαση. Ε, ε, υπάρχει και μια διαφορετική μεθοδολογία όταν σε προηγούμενες εκλογές ήταν παρούσα μια αντιπροσωπεία παρατήρησης εκλογών δήλωσε ότι υπήρξαν ελλείψεις και μειονεκτήματα στην εκλογική διαδικασία. Αν εμείς τώρα κληθούμε να παρευρεθούμε και αν αντιμετωπίσουμε συγκεκριμένες ελλείψεις κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, αν διαπιστώσουμε ελλείψεις, θα πρέπει να περιμένουμε, όπως έλεγα στον κύριο Πίμπαλ προηγουμένως, Λέτε ότι έχουμε ρόλο διαιτητών. Φανταστείτε ένα διαιτητή που δεν μπορεί να σφυρίξει παρά μόνο όταν τελειώσει ο αγώνα. Γιατί σε τέτοια κατάσταση μπαίνουμε. Μα λένε ότι εμεί είμαστε οι διαιτητέ, αλλά δεν μπορούμε να παρέμβουμε καθόλου. κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του αγώνα ο διαιτητής δεν μπορεί να παρέμβει γιατί θα θεωρηθεί παρέμβαση αυτό. Είναι τόσο κέρια σημασία στα διακυβεύματα εδώ που βλέπουμε ότι οποιαδήποτε έλλειψη μπορεί να οδηγήσει και σε βία. Επομένως πρέπει να δούμε κατά πόσο μπορούμε να παρέμβουμε και πώς με τρόπο διακριτικό, ίσως όχι με ανοιχτό τρόπο, αλλά πώς μπορούμε να προσπαθήσουμε να διορθώσουμε τις ατέλειες που βλέπουμε, ώστε να μην φτάσουμε στο τέλος σε μια έκθεση για την αποστολή μας στις εκλογές που θα δημιουργήσει εκρηκτικές αντιδράσεις. Θα πούμε κάνατε το τάδε το τάδε σφάλμα και θα μας πούμε γιατί δεν μας το είπατε όταν θα μπορούσαμε να παρέμβουμε. Όλα αυτά τα θέματα λοιπόν τίθενται σήμερα ως ερωτήματα για το μέλλον του Σουδάν. Και εγώ μίλησα μόνο για τα τεχνικά θέματα που αντιμετωπίσαμε στην ε, αποστολή παρατήρηση των εκλογών. Η έκθεση που υποβάλαμε ήταν δύσκολη να την αποδεχθούν οι Σουδανοί, γιατί τους είπα ότι ε, βγάλατε αποτελέσματα με λιγότερο το 50%, ε, αλλά όταν το έλαβαν το μήνυμα έδειξαν πολιτική οριμότητα. Ε, υπήρχε μια εσωτερική διαμάχη με την Επιτροπή των Εκλογών, που δεν θα είναι όμως η Επιτροπή του Δημοψηφίσματος, και η κυβέρνηση στο Βορρά δέχθηκε το μήνυμα που τους δώσαμε και είπαν ναι, πρέπει να, να βγάλουμε τα συμπεράσματα για το μέλλον, να προσέξουμε τι θα γίνει στο δημοψήφισμα και το ίδιο πρέπει να γίνει και στο Νότο. Και το αυτό ήταν πολύ θετικό. Είπαν ε, ε, πολλοί ότι ήταν πρώτη φορά που ψηφίζουμε εδώ και πάνω από 20 χρόνια. Αυτές οι εκλογές ήταν πάρα πολύ ε, πολύπλοκες. Είχαμε 12 ψηφοδέλτια, νομοθετικές, προεδρικές κλπ. Πάρα πολλές εκλογές, πολύ πολύπλοκα. Θα τα καταφέρουμε καλύτερα την επόμενη φορά. Το αναγνώρισαν λοιπόν. Αυτά για να κλείσουμε κάπως θετική νότα. Ευχαριστούμε. Και τώρα θα ζητήσω την κυρία Γκόμες να λάβει το λόγο ήταν πρόεδρος της δικής μας κοινοβουλευτικής ομάδας παρατηρητών. Αλλά θα σας παρακαλέσω, επειδή έχουμε ακόμη πέντε αγορητές μετά από εσάς και θα πρέπει να τεθούν ερωτήματα και να δοθούν και απαντήσεις. Και ξέρετε ότι στις 6.30 θα φύγουν και οι άνθρωποι από τις καμπίνες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρέπει να πω ότι συμφωνώ απολύτως με όσο είπε η και με τις προειδοποίησεις που εξέφρασε, ιδίω για την οργάνωση του δημοψηφίσματος τον Ιανουάριο. Υπάρχει ανάγκη παρέμβαση στην κατάλληλη στιγμή. Και νομίζω στο πλαίσιο των κατευθυντηρίων γραμμών μας, των συστάσεών μας, θα πρέπει να υπάρχει κάποιο περιθώριο να μπορούμε να σφυρίξουμε σαν διαιτητές την κατάλληλη στιγμή και όχι εκ των υστέρων. Εάν παίρνουμε σοβαρά το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μάλιστα, των και όλες, όλα αυτά τα θέματα που θα πρέπει να τηρούνται κατά τη διάρκεια της εξαγωγής εκλογών αν θέλουμε να είναι Εγώ για την αποστολή αυτή στο Σουδάν είχα δικαιολογημένη παρουσία και είχα και πολλές προκαταλήψεις πριν πάω αλλά άλλαξε η άποψή μου όταν μετέβηνε επί τόπου γνώρισα καλύτερα τι συμβαίνει στο Σουδάν και μπορεί κανεί έτσι, κανείς έτσι να προετοιμαστεί καλύτερα και για το μέλλον και μάλιστα και στο περιθώριο του δημοψηφίσματο. Να πω ότι τα μαθήματα που θα πρέπει να συγκρατήσουμε για το μέλλον, για το δημοψήφισμα, όπως πολύ σωστά τα επεσήμανε και η Βερονίκ, είναι ότι υπάρχει πραγματικός κίνδυνος να οδηγηθούμε σε άλλη δικτατορία ή σε άλλο κράτος ε, ανεξάρτητο. Εδώ, από πλευρά Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν μιλάμε μόνο για την εκλογική προετοιμασία, που είναι ένα σημαντικό μέρο τη όλη διαδικασία. Στον Βορρά, οι εκλογέ αυτέ απέδειξαν ότι δεν μπορούμε να παραβλέπουμε την δημοκρατική μετατροπή του Σουδάν, ιδίω, στο Βορρά, οι πολίτες έχουν λάβει το μήνυμα αυτό και θέλουν να το δώσουν να το καταλάβουμε, ότι θέλουν να αλλάξει η χώρα. Υπήρξαν και αυταρχικέ δηλώσεις του Πρόεδρου Μπασίρ πριν τι εκλογές, εξαπειλούσε απειλέ ότι θα κόψει γλώσσες και δάχτυλα για, τις, ε, για το ενδεχόμενο αναβολή εκλογών. Αλλά αντιθέτως με το ότι περιμέναμε, μας καλωσόρισαν στο Σουδάν. Μας είπαν πόσο καταδίκαζαν έντονα τις δηλώσεις του Πρόεδρου Μπασίρ. Και στη συμπεριφορά τους και στην υποδοχή μας επεφύλαξαν πραγματικά στο βορρά, στους ανθρώπους του. Είδαμε ήδη μέσα σε πέντε μέρες τις πέντε μέρες των, της δεξαγωγής των εκλογών ότι υπήρχαν πολλά κενά βεβαίως, υπήρχαν αδυναμίες, αλλά όχι μόνο με το κυβερνόν κόμμα. Όλοι όσοι συμμετείχαν φαίνεται να θεωρούν δεδομένο ότι το κυβερνόν κόμμα μπορούσε να λάβει ένα πλήρη κατάλογο με τους ψηφίσαντες και να πάνε στα διάφορα σπίτια και να να πούνε στου εκλογέ τι πρέπει να ψηφίσουν. Αλλά αυτές οι απόψεις μπορεί να ασκηθεί και να αλλάξουν και γίνονται όλε οι απαραίτητε προσπάθειε. Είναι επίση σημαντικό να μην παραβλέπουμε τον Ταρφούρ. Και πάλι στηρίζω την απόφαση της Βερονίκ, νομίζω ότι ήταν σοφή και δεν νομίζω ότι έγινε κατανοητή από την ε, πρόσωπο της Επιτροπής, της Επιτροπής την κυρία Άστον. Σωστά ε, είπε η Βερονίκο ότι δεν γινόταν να διοργανωθεί παρατήρηση των εκλογών στον Ταρφούρ, έκανε εκλογέ δεν γινόταν να διοργανωθούν εκεί. Τα προβλήματα εκεί ήταν ακόμη χειρότερα. Ε, με τους ανθρώπους που ήταν απομονωμένοι στους καταπλησμούς. Τέλος, δεν πρέπει να ξεχνούμε το τι έγινε στο δαρφούρ μετά. Τα πράγματα επιδεινώθηκαν. Οι νευτικές συνομιλίες δεν οδηγούν πουθενά. Και υπήρξαν και αρνητικές εξελίξεις με την ε, σύλληψη του βασικού αντιπάλου του πρόεδρου Μπασίρ. Και ο κύριος Μαχμούτος Μαντ και εκείνο και τα μέλη της αντιπροσωπεία τη μη κυβερνητική Οργάνωση δεν μπορούσαν να πάνε στην ε, συνεδρία αναθεώρηση τη Καμπάλα, τη ΑΕΣΥΣ. E δεν είχε θεώρηση για να μεταβεί και μόλι το επιστράφει. Ο το του. Θα πρέπει λοιπόν να παραμείνουμε προσεκτικοί στην παρατήρηση των εκλογών. Ο κύριος Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, χαίρομαι ιδιαίτερα διότι ο πρέσβης, ε, ο κύριος Μπρίλε, ήρθε ε, τόσο σύντομα να μας επισκεφθεί στην Επιτροπή μας. Ειδωθήκαμε το Μάιο στο Χαρτούμ, δεν είμαι ειδικό όπως η κυρία Γκόμες, η κυρία Ντεκάιζερ, αλλά μετέβη και εγώ μονομένα στο Χαρτούμ και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά τα οποία ε, ε, μας είπατε σε σχέση με την κατάσταση αυτή. Έχω κάποιες συγκεκριμένες ερωτήσεις. Δεν ξέρω πώς να το εκφράσω. Κάπως ανησύχησα γιατί και πάλι ε, συζητήσατε όπως και στα τέλη Μαΐου που συναντηθήκαμε στο Χαρτούμ είπατε τώρα ότι δεν υπάρχει οριοθέτηση των συνόρων. Είναι σημαντικό να οριοθετηθεί η εκλογική περιφέρεια. Μας ενδιαφέρει λοιπόν να δούμε ποιες είναι οι μέθοδοι βάσει των οποίων ε, θα οριοθετηθεί η περιοχή στις οποίες θα γίνουν εκλογές και ποιοι είναι οι διεθνείς φορείς, τα Ηνωμένα Έθνη, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, η Ρωσία, ποιοι θα συμμετάσχουν σε αυτή τη διαδικασία για να γίνει αυτή η οριοθέτηση. Γιατί χωρίς να γίνει η οριοθέτηση, το να φτάσουμε στο δημοψήφισμα, κατά τη γνώμη μου θα είναι πολύ επικίνδυνο. Ευχαριστούμε κύριο Στάνοκ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Εγώ συμμερίζομαι την άποψη της Άννας Γκόμες. Δεν ξέρω αν ήταν συνετό να αποσταλεί τέτοια παρατήρηση υψηλού επίπεδου για εκλογές ενώ ένας από τους υποψηφίους ήταν ένας καταδικασμένος ε, εγκληματής πολέμου για γενοκτονία όπως πρόσφατα ανακοινώθηκε από τον εισαγγελέα του ενδιάμεσου ποινικού δικαστηρίου, του προσωρινού ποινικού δικαστηρίου, συγγνώμη. Πάντως φαίνεται να ήταν αυτό μια γενική πρόβα για τις πολύ σημαντικότερες εκλογές της επόμενης χρονιάς, για την ανεξαρτησία του Νότου. Αύριο μάλιστα θα οργανωθεί γεύμα με τον κύριο Πέγκαν και έναν από τους υπουργού του Νότου, όπου θα είμαι εγώ υπεύθυνο για την φιλοξενία και να συζητήσουμε για τα θέματα αυτά και να δούμε τις συνομιλίες που μπορούμε να έχουμε με τους υποστηρικτέ μεταξύ των βουλευτών. Τώρα, όσο τα πράγματα εντείνονται μεταξύ Βορρά και Νότου, πιστεύετε ότι εδώ θα μπορούσε να έχουμε έναν εισαγόμενο πόλεμο που να σχετιστεί με τη λαϊκή δημοκρατία της Κίνας και το επίσημο καθεστώς του πρόεδρου Μπασίρ στο Χαρτούμ αλλά και μεταξύ των Πολιτείων που ασκούν πιέσεις στο Κογκρέσο. Χριστιανικό κύριος ε, λόμπι για την ανεξαρτησία του Νότου. Πιστεύετε ότι μπορεί να αναπτυχθούν λοιπόν ε, κατ' επέκταση εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας εάν υπάρξει ενίσχυση του αποσχιστικού κινήματος του Νότου και πιστεύετε ότι θα ληφθούν μέτρα για, από την πλευρά του Βορρά για τον έλεγχο του Νότου ή θα παραμείνει ουδέτερος. Και επίσης την περασμένη εβδομάδα είδαμε ότι στην περιοχή της Σομαλίας που αποσχίστηκε Στη Σομάλιλαντ είχαμε ανεξάρτητες και αδιάβλητες εκλογές. Θα πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε στο Νότο να δούμε κατά πόσον μπορούν να γίνουν αντακειμενικές εκλογές. Δεν θα πρέπει να ακολουθεί το παράδειγμα της Σομάλιλαντ και εκεί. Ευχαριστούμε κυρία Λέζιν. Ähm, Ευχαριστώ πολύ. Οι συζητήσεις για το μέλλον έχουν κάπως ε, τροποποιηθεί και ε, προσφάτως συζητήσατε και με τον Τάμπο Μπέκη, με τον οποίο και εμείς είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε ε, κάποια στιγμή. Ανέφερε προσφάτως κάτι για συνομοσπονδία, έφερε την ιδέα της συνομοσπονδίας στη συζήτηση και εκφράστηκε υπέρ αυτής της άποψης ε, και μέσα στο SPLM ε, υπήρξαν αντιθέσεις. Αν ε, λοιπόν δούμε πώς έχει η κατάσταση αυτή τη στιγμή και βλέπουμε ότι οι πόροι είναι άνισα καταναμημένοι στα δύο τμήματα της χώρας, ο Βορράς δεν είναι σε καλή κατάσταση όσον αφορά τους πόρους και από γεωργικής ε, ε, παραγωγή, από γεωργικής παραγωγής, αλλά και οι πετρελαϊκοί πόροι βρίσκονται ε, στο νότο. 5 δισεκατομμύρια βαρέλια, η τέταρτη υψηλότερη το τέταρτο υψηλότερο δυναμικό της Αφρικής βρίσκεται στο Σουδάν. Τίθεται λοιπόν εύλογα το ερώτημα πόσο θετική θα είναι η απόσχηση του Νότου για μια μελλοντική βιώσιμη ειρήνη. Και ίσως είναι κάτι το οποίο δεν βασίζεται σε παραδοσιακές απόψεις. Ο Τζον Γκάραν ε, δεν υπάρχει πια και ε, θα πρέπει να δούμε ποια είναι τα επιχειρήματα υπέρ. Πρέπει επίσης να πούμε ότι ε, και από την πλευρά του SPLMA υπάρχουν ε, επιθέσεις κατά των ε, αντιπάλων, άρα υπάρχουν αντίστοιχη κατάσταση και στο Νότο δεν ξέρω λοιπόν αν μπορούμε να υποστηρίζουμε την απόσχεση του Νότου στη Δύση. Αυτή είναι η ερώτησή μου λοιπόν, ε, εάν πολιτικά έχει νόημα το να κινηθούμε προς μια συνομοσπονδία. και κατά αυτόν τον τρόπο η ενότητα του Σουδάν θα είναι κάτι το οποίο θα παρουσιάζεται ε, πιο ελκυστικά προς τους πολίτες ε, του Νότου, του Σουδάν. Ε, και μια συγκεκριμένη ερώτηση πόση βοήθεια δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο Βορρά και πόση στο Νότο. Και όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, ε, σας είπα ότι το SPLMA ε, έχει επίσης ε, κάνει επιθέσεις που πρέπει να αναφέρονται. και υπάρχουν και περιπτώσει στρατιωτική υποστήριξη. Θα ήθελα να ακούσω τα σχόλιά σα από αυτού και τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να ασκήσει πίεση στο SPLM να τηρήσει τα δικαιώματα ε, των αντιπάλων του. Ευχαριστώ πολύ. Κύριο Σαγκουράκης, παρακαλώ. Ε, και σκεφτείτε και το χρόνο. Ε, θα συνεχίσω στα ελληνικά. από την παρέμβαση του κυρίου Πρέσβη όσον αφορά το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος κατάλαβα ότι λίγο πολύ προεξοφλεί το αποτέλεσμα. Μας είπε ο κύριος Πρέσβης, αν ε, καλά κατάλαβα, αυτό μεταφράστηκε, ότι ανεξάρτητα ποιο θα είναι το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος, αυτό που απασχολεί είναι η μέρα μετά. Και στη μέρα μετά αναφέρθηκε σε τέτοια προβλήματα που αφορούν δύο ανεξάρτητα κράτη. Δηλαδή προεξοφλούμε από τώρα ότι το δημοψήφισμα θα είναι υπέρ της ανεξαρτησίας του, ε, του Νότου. Ένα ερώτημα είναι αυτό. Ε, δεύτερο ερώτημα. Ε, στις εκλογές που γίναν πρόσφατα στο Σουδάν, το θέμα του δημοψηφίσματος και της ανεξαρτησίας του Νότου ήταν θέμα στις εκλογές, στο Βορρά, παντού. Ποια είναι η γενική άποψη που υπάρχει. Τρίτο ζήτημα, και εγώ θα συμφωνήσω με την κυρία Λέζινγκ, δεν θεωρώ το θέμα της ανεξαρτησίας λύσης. Από ό,τι γνωρίζω, βασικός παράγοντας σε αυτή την επιλογή είναι το πετρέλαιο, που είναι συγκεντρωμένο στο νότιο τμήμα της χώρας και για το πετρέλαιο, όπως γνωρίζουμε, γίνονται πολλά και διάφορα αυτή την εποχή. Ε, θα ήθελα ωστόσο να ε, σημειώσω το εξής ε, ζήτημα. Στην περίπτωση που θα γίνει το δημοψήφισμα, ποιος θα το οργανώσει το δημοψήφισμα, ποιο, ποιος θα είναι ο φορέας που θα το οργανώσει εκ μέρους των Σουδανών, όχι η διεθνής κοινότητα, ο ΙΕ, ε, η Αφρικανική Ένωση. Και τελειώνοντας, επειδή έγινε λόγος για τον διαιτητή, ε, σε αυτά τα ζητήματα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Εάν σκοπεύουμε να παρέμβουμε στις εκλογές, όπως υπόθηκε, να αναλάβουμε όμως και τις ευθύνες ως Ευρωπαϊκή Ένωση το τι θα ακολουθήσει μετά από μια τέτοια παρέμβαση. Γι' αυτό νομίζω είναι πολύ σημαντικό να ξεχωρίσει κανείς το ρόλο του παρατηρητή από του ρόλου αυτού που κάνει τις εκλογές. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ, ο κύριος Βάγγελ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εξοχότατε, κύριε ε, Πρέσβη. Δεν θα μπω στον πειρασμό να συμφωνήσω με τους συναδέλφους που μίλησαν για ε, το πρόβλημα του Νότου και το, το, πρόβλημα του Σουδάν γενικά. Θα μιλήσω για τον Ταρφούρ μόνο και τις διαπραγματεύσεις της Ντόχα. Εσείς πώς εξετάζετε και πώς αξιολογείτε αυτό το θέμα. Έχουν ε, πεθάνει πλέον οι διαπραγματεύσεις. Ήρθε εδώ ο κύριος Σουλεμάν Τζομούς, το γνωρίζετε με βέβαιος, και εξέφρασε τα παράπονα ότι στην Τόχα, στο Κατάρ, το πρόβλημα στις διαπραγματεύσεις ήταν ότι υπήρχαν κάποιοι υποτιθέμενοι οργανισμοί της κοινωνίας των πολιτών που είχαν δημιουργηθεί τεχνητά απλώς και μόνο για να αυξηθεί ο αριθμός των ε, συμμετεχόντων και να θολώσουν τα νερά και να ε, αποσπάσουν την προσοχή από τις πραγματικές οργανώσεις που έπρεπε να έχουν λόγο και να εκπροσωπούν το λαό. Σας ερωτώ λοιπόν τι πιστεύετε για την Τόχα και τι για τον Νταρφούρ. Γίνεται τίποτα εκεί, κινείται τίποτα. Γιατί προφανώς αν στο νότιο Σουδάν διακυβεύεται το πετρέλαιο, στο Νταρφούρ διακυβεύεται το νερό. Ξέρετε τι έγινε τις περίσμενες εβδομάδες στη Τζάμπελ Μάρα. Ε, αυτά μιλούν από μόνα τους. είναι φίλιος πόλεμος και η γενοκτονία που θα επιδεινωθεί διότι εκεί πραγματικά δεν τσακώνεται για το πετρέλαιο αλλά για το νερό. Ευχαριστώ. Κύριε Πρέσβη, έχετε το λόγο. Γιατί ε, τέθησαν και θέματα παρατήρησης εκλογών. Θα ζητήσω το τέλος τη Βερονίκη να συνοψίσει. Ευχαριστώ, ευχαριστώ όλους για τις παρεμβάσεις σας και τις ερωτήσεις σας. Πρώτα απ' όλα να απαντήσω για το ζήτημα που έθεσε ο κ. Πέτερη. Ναι, με την άποψη ότι η μη καλή οριοθέτηση των σύνορων στον Νότο είναι σημαντικό πρόβλημα. Είχα ευκαιρίε σήμερα να συζητήσω την κατάσταση του Σουδάν με τον Υπουργό Πακανεμούν, ο οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην κυβέρνηση του Νοτιού Σουδάν για την ειρήνη και την συμμετοχή στην ολοκληρωμένη συμφωνία ειρήνευσης και επιβεβαίωσε ότι και για τους ίδιους το ζήτημα αυτό είναι κέρια σημασία. Όλοι καταλαβαίνουν ότι αν κανείς δεν είναι βέβαιος που βρίσκονται τα σύνορά του, μόνο σε συνθήκε αβεβαιότητας μπορεί να ζει. Αυτό που συμφωνήθηκε είναι το 80% περίπου των σύνορων, όμως το υπόλοιπο 20% είναι κρεμή ζητήματα και φαίνεται να υπάρχει τέλμα στο επίπεδο τη επιτροπή και στην εξέταση του ζητήματο αυτού. Ξέρω ότι απευθύνθηκε έκκληση για διεθνή στήριξη, τεχνική στήριξη από την ε, αποστολή για την ε, ενδιάμεση, ε, για την ολοκληρωμένη ειρηνευτική συμφωνία για το θέμα αυτό. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε λοιπόν από πλευρά διεθνού κοινότητα για να παράσχουμε τεχνική στήριξη ω προ την... του διεθνεί ενδιαφερομένου και την αποτίμησή τους και την δεσμευσή τους και την προσέγγιση προς το Σουδάν, νομίζω ότι υπάρχει μια τάση σύγκλησης εδώ. Υπάρχει γενικώ αναγνώριση ότι έχουμε περάσει στην αντίστροφη μέτρηση προς μια κρίσιμη στιγμή. Έχουμε μια ενδιάμεση περίοδο μέχρι την κρίσιμη αυτή στιγμή και θα φανεί πώς θα, τι στάση θα κρατήσει πλέον το Σουδάν, άσχετα με το τι δρόμο θα πάρει ο Νότος. Θα δούμε αν μπορεί να υπάρξει ειρηνική συνύπαρξη. Υπάρχει απόκληση απόψεων βεβαίω. Υπάρχουν ε, διαφορετικέ απόψεις. αλλά όλοι συμφωνούν στο ότι πρέπει η κατάσταση να υποφελήσει και τις δύο πλευρές. Επίση, στο επίπεδο των διεθνών μα ε, συναντήσεων, των διαλόγων που έχουμε σε πολλές ε, περιπτώσεις δεν έχουμε όλοι ακριβώς τις ίδιες απόψεις, όμως παγκοσμίω υπάρχει συμφωνία. Πρέπει να εργαστούμε για την ειρήνη και τη σταθερότητα στο Σουδάν. Εγώ δεν βλέπω πρόπτικη να υπάρξει ένας ε, εισαγόμενος πόλεμος μεταξύ των ε, μεγάλων δυνάμεων του πλανήτη στο Σουδάν. Δεν υπάρχει βεβαίω αρκετή σταθερότητα ακόμη στο Σουδάν, υπάρχουν αντικρώμενα συμφέροντα. Όμω όλοι θέλουν να λάβουν τι ευθύνε του και όλοι να γνωρίζουν ότι η κατάσταση είναι ιδιαίτερα περίπλοκη. Και ότι μπορεί να επιληθεί μόνο με όρου πολιτικού το πρόβλημα. Επίση ερωτήθηκα για το ρόλο του πρώην Προέδρου Εμπίκη που ορίστηκε από την πρώην Αφρικανική Ένωση στο αρμόδιο πάνελ. Θεωρούνται διευκολυντές και, χρησιμοποιούν το μνημόνιο συνεννόησης Μακέλη ως διαπραγματευτικό αντικείμενο. Υπάρχουν και εδώ διαφορετικέ απόψει για το πώ μπορεί να εξακολουθήσει η ειρηνική συνύπαρξη στο ερχόμενο διάστημα. Εδώ νομίζω υπάρχει επίση συνένεση. Όπω συχνά συμβαίνει σε τέτοιε περιπτώσει στην Αφρική, εδώ είναι ε, ένας βασικός λόγος για τη σύγκρουση, η φυσική πόρη. Στην περίπτωση του Σουδάν και πάλι αυτό εκτός από αφορμή σύγκρουση μπορεί να γίνει και ευκαιρία διότι το πετρέλαιο μπορεί να φεύγει από τον νότο προς το βορρά και αυτή να είναι η δίωδος προς τα έξω. Υπάρχουν λοιπόν αμοιβαία συμφέροντα για τη διαχείριση των φυσικών πόρων στο Σουδάν. Και αυτό που εγώ και τι δύο πλευρέ είναι ότι κατανοούν και οι μεν και οι δε ότι είναι ιστορικά δεμένοι μεταξύ του. Υπάρχουν άνθρωποι από το βορρά που ζουν στο νότο και αντιστρόφω. Η διαβίωσή του είναι... εξαρτάται. Η διαβίωση του ενό από το πώ ζει ο άλλο. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχουν σχέσει εμπιστοσύνη μεταξύ των πλευρών, κάτι που δεν υπάρχει ακόμη, όμω καταλαβαίνουν ότι οι μεν έχουν ανάγκη του δε και πρέπει να εξεύρουν συστήματα που να υποφελούν και τους δύο. Το 2005 όταν συνήθη η συμφωνία, η ολοκληρωμένη συμφωνία, η ειρηνευτική συμφωνία και οι δύο πλευρές αναγνώρισαν την ανάγκη να πάψει ο πόλεμος και αυτό ισχύει ακόμη. Ε, ήταν ελκυστική, ελκυστικό το όραμα που είχαν ήδη συλλάβει όσοι επεξεργάστηκαν την συμφωνία αυτή, την Ειρηνευτική Συμφωνία του 2005 και αυτό ίσχυε ακόμη. Την επεξεργάστηκαν οι ηγέτες του Νότου και δεν ισχύουν βέβαια όλα τα πράγματα με τον ίδιο τρόπο, όμως ε, θα πρέπει να αφήσουμε τους ίδιους να αποφασίσουν. Δεν μπορούμε να προδικάσουμε κανένα αποτέλεσμα. Υπάρχει ανάγκη στήριξης εδώ, αναπτυξιακής δηλαδή στήριξης, προς όλες τις κατευθύνσεις, όχι μόνο προς τον Νότιο Σουδάν. Προβλέπεται μάλιστα ένα κονδύλι 50 εκατομμυρίων ευρώ της PNL για τους πληγέντες από τον πόλεμο. Γκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή χθε νομίζω. Και ίσως έθιξε το θέμα του πετρελαίου και των φυσικών πόρων. Τώρα για το ποιος θα διοργανώσει το δημοψήφισμα. Αυτό το αναλαμβάνει η Επιτροπή Δημοψηφίσματος, η οποία πρόσφατα διορίστηκε. Και όπως και με τις εκλογές που ανατέθηκαν, στα χέρια της αρμόδιας εκλογικής επιτροπής, η Επιτροπή του Δημοψηφίσματος είναι εκείνη που θα αναλάβει. Είναι ανεξάρτητο σώμα με τεχνική αρμοδιότητα και ο ΙΕ θα διασφαλίσει τη λειτουργία του, αλλά σίγουρα θα διοργανωθεί καταλήλως. Τώρα για τον Ταρφούρ και το θέμα της πολιτικής διαδικασίας. Νομίζω ότι κάλυψε το θέμα του Νταρφούρ. Υπάρχει θέμα ασφαλείας, ιδίως στο νότιο Νταρφούρ. Οι δυνάμει στήριξη τη ειρήνη ε, δυσκολεύονται να πληρώσουν την αποστολή του προ την προστασία των αμάχων και την ε, βασική ασφάλεια. Υπάρχει δυσκολία πρόσβαση και των ε, δυνάμεων αυτών και των διαπραγματευτών και βεβαίω υπάρχουν βαθιέ ανησυχίε από όλες τις πλευρές ότι ε, η δολοφονία των ε, μελών της ειρηνευτικής αποστολής είναι έγκλημα πολέμου βεβαίως. Έτσι καταλαβαίνουμε γιατί υπάρχει αρνητικός αντίκτυπο στο κατά πόσο μπορεί να παρασχεθεί ανθρωπιστική βοήθεια. Υπάρχει επίσης ε, συνυπευθυνότητα του Χαρτούμ και το υπεσήμενα αυτό στον Υπουργό Ανθρωπιστικών Υποθέσεων στο Χαρτούμ που μου είπε ότι τα σχετικά ζητήματα τα εξετάζει, εξετάζει όλο τον κατάλογο των σχετικών ζητημάτων και τον ερχόμενο μήνα θα συζητήσει σε ανώτερο επίπεδο τα θέματα αυτά. Είναι πολύ σημαντικά για όλους στον Τερφούρ. Τώρα η πολιτική διαδικασία στην Τόχα είναι ακόμη ζωντανή. Υπάρχουν συζητήσεις μεταξύ κυβερνήσεων, συνασπισμών, πολιτικών. Την ώρα που μιλάμε, μόλις χθες είχαμε τα εγγένεια ενό φόρουμ τη Κοινωνία των πολιτών. 450 ε, πολίτε συμμετέχουν εκεί. Δεν ξέρω τώρα αν είναι πραγματικά πολίτες απλοί, αλλά κάτι διαφορετικό θα ήταν περίεργο δεδομένη τη κατάσταση των Ταρφούρ. Εμεί είμαστε μεταξύ όσων συνηγόρησαν υπέρ τη ανάγκη συμμετοχή τη κοινωνία των πολιτών, ώστε οι φωνέ των πολιτών να ακουστούν. Και αυτό θα συνεχίσουμε να το υποστηρίζουμε. Βεβαίω υπάρχει περιορισμένο αριθμό ε, καθισμάτων γύρω από το διαπραγματευτικό τραπέζι. Όμω, ακόμη και αν όλοι αυτοί δεν συμμετάσχουν στι διαπραγματεύσει, μπορούν τουλάχιστον να δεδοθούν ότι θα τεθούν επιτάπητο οι ανησυχίε του. Για να καταφέρουμε συμφωνίε διαρκεία κατά αυτόν τον τρόπο. Η Ντόχα δεν είναι η τελεσίδικη, οριστική επίλυση και δυνατότητα συμμετοχή τη κοινωνία των πολιτών. Όσοι έχουν ασχοληθεί με το κίνημα ισότητα και ελευθερίας ξέρουν ότι ε, προσπαθούμε να τους ε, φέρουμε ε, σε διαπραγματεύσεις. Δεν τους έχουμε πείσει ακόμη, προσπαθούμε, αλλά ωστόσο ο στόχος είναι να τους εξηγήσουμε ότι είναι προς όφελός τους. Και έτσι η συμφωνία της Αβούτζα από το 2006 μπορεί να οδηγήσει στο να μεταλλάξουν τη στάση τους και για τον τερφούρ και πολύ από τον τερφούρ. Ελπίζω, ελπίζω ότι κάλυψα τα ζητήματα που τέθηκαν. Ε, αυτή ήταν τουλάχιστον η πρόθεσή μου, εάν υπάρχουν να Βερονίκ, θέλεις να πεις τίποτα για όλα αυτά. Έχεις δύο λεπτά. Το πολύ. Chercher où Πάρα πολύ σύντομα. Για το ποιος διοργανώνει τις εκλογές. Είναι σαφές και έχει δίκιο ο συνάδελφος να το λέει. Είναι η ιδανική κυβέρνηση και αυτή θα πρέπει να ελέγχει και τις εκλογές. Όταν είπα αν χρειαστεί να παρεύουμε, όχι για να επέβουμε, να αναμειχθούμε στα εσωτερικά της χώρας, γύρω από τη Σουδανική κυβέρνηση και τη Φορευτική Επιτροπή χρειάζεται κάποια πλαισίωση, κάποια υποστήριξη. Η υποστήριξη του ΟΗΕ, πούμε, για τη διοργάνωση, ε, την επιμελητία των εκλογών. Επίσης, ήτανε ε, ακριβώς η προετοιμασία για το λογισμικό, όλα τα τεχνικά ζητήματα. Είμαστε εκεί ε, μόνο υποστηρικτικά. Η ε, εκλογική παρατήρηση θα πρέπει να είναι απαλλαγμένη από όλα αυτά και να παρατηρεί μόνο τις εκλογές και τίποτα άλλο. Αλλά συχνά υπάρχουν κανόνες που διαφέρουν πάρα πολύ για την παρατήρηση. Το κέντρο του Κάρτερ ανησύχησε για τον τρόπο με τον οποίο γινόταν η εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους. Και ξέρω ότι ο Κάρτερ είχε πάει στον πρόεδρο Αλμπασίρη και συναντήθηκε μαζί του και μετά αφού είδαν ε, ότι υπήρξε νοθεία ε, η παραβίαση των προτύπων έβγαλε μια ενδιάμεση έκθεση και εξέφρασε τη δυσφορία του, εν πάση περιπτώσει, για ορισμένες καταστάσεις και ζητούσε ε, σε άλλη ενδιάμεση έκθεση να αναβληθούν οι εκλογές διότι δεν ήταν ε, ακόμα έτοιμοι. Δηλαδή είχε κάποιες μικρές παρεμβάσεις ο Κάρτερ και ο Αλμπασίρ, ο πρόεδρος του Σουντάν, το πήρε πολύ άσχημα γιατί έκανε δύο ε, ομιλίες αρκετά εμπριστικές και είπε ότι ναι θα σας κόψουμε τα πάντα, τα χέρια, τα πόδια, ε, τα δάχτυλα, τις μύτες, ε, αν θα αναπηγνιόμασταν και ανησύχησαν οι παρατηρητές γιατί δεν περίμενε ο πρόεδρος χώρας να πει τέτοια πράγματα. Αλλά όταν είμαστε σε μια τέτοια χώρα τόσο μεγάλη όσο Ήπειρος, ε, μπορεί κάποιοι τρελοί να το πάρουν και τις μετρητές και να αρχίσουν να κόβουν. Ε, δηλαδή φοβηθήκαμε, θορυβηθήκαμε λίγο. δεν σημαίνει ότι γι' αυτό θα πρέπει να προσέχουμε, πάντα θα πρέπει να προσέχουμε. Εγώ δεν αρνήθηκα ποτέ ε, κάτι τέτοιο, αλλά θα πρέπει να δούμε πώς θα βοηθήσουμε καλύτερα μια χώρα που μπαίνει σε μια περιπέτεια τόσο σημαντική και χρειάζεται υποστήριξη. Και ένα δεύτερο που θα ήθελα να αναφέρω από όλε τι συνομιλίε και τι επαφέ που είχα στο Σουντά, μπορώ να σα πω ότι στο Νότο, αν μη τι άλλο, δεν ευσταθεί πλέον η ιδέα τη ενιαία χώρα. Το λένε στα αγγλικά αυτό too little and too late, πολύ λίγα και πολύ αργά έρχονται από το βορρά και τους λένε πώς θα μοιραστούν τους πλουτοπαραγωγικούς πόρους, πώς θα γίνει δίκαιη κατανομή, γιατί ε, βασικά ο πλούτος είναι γύρω από τη χαρτούμ, ούτε ο, ο βορράς, ο πόλτος, ούτε ο νότος είναι ανεπτυγμένοι. Τώρα υποτίθεται ότι γίνονται κάποιες προσπάθειες, αλλά είναι πάρα πολύ λίγα αυτά και πάρα πολύ αργά. Είναι μια υπανάπτυξη διαδεδομένη σε όλη την περιφέρεια του Σουδάν και έχει διατηρηθεί εσκεμένα σε αυτή την κατάσταση και καθόλου δεν είναι ελκυστική η ιδέα της ενιαίας χώρας για τον Νότο. Και περιέργως οι Νότιοι Σουδανοί λένε με πολύ μεγάλη σοβαρότητα ότι αν τι άλλο όχι τώρα. Δηλαδή όσο κυβερνάει ο πρόεδρος Αλ Μπασίρ ε, προτιμούμε να τηρήσουμε τις αποστάσεις μας. Θα δούμε μετά μήπως χρειαστεί να επανενωθούμε δεν είναι περίεργο, δηλαδή ότι προσωρινά αποσχιστούμε και μπορεί αργότερα να τα ξαναφτιάξουμε και να κάνουμε ενιαία χώρα. Το λένε αυτό και το λένε και σοβαρά πολύ στο Νότιο Σουδάν. Αρκετά περίεργο είναι όμως έτσι ως ε, συλλογισμός. Και τέλος, αν υπάρχει ένα σημείο που ήταν σημαντικό για τη δημοκρατία, ένα και μόνο, στις εκλογές αυτές ήταν ή εγχώριοι παρατηρητές και η κατάρτισή τους. Αυτό λέγεται domestic observers. Αυτή είναι η κοινωνία των πολιτών που ανησυχούν, που γνωρίζουν, ε, από πολλού και το κέντρο Κάρτερ ακριβώς έκανε πολύ μεγάλη δουλειά εκεί στην κατάρτιση. Είναι μια στοιχειώδης κοινωνία των πολιτών ε, που έχουν όμως το κάθε, κάθε κύρος να ασχολούνται με τις εκλογές είναι νέοι, πάρα πολύ ικανοί, με πάρα πολλά εφόδια και ελπίδα για το μέλλον του Σουδάν. Αυτά, τελείωσα, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Πρέσβη, θα σας ευχαριστώ όλους σας. Κάνετε πολύ καλή δουλειά.